Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die Sitzung. Zunächst äh, möchte ich... Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις για την παρουσία της ε, ε δεύτερης γερμανικής ε, δημόσιας τηλεόρασης εδώ, η οποία θα φιλμάρει. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Έχετε όλη την ημερησία διάταξη λοιπόν. Ο κύριος, κύριος Σόλτς θα ήθελε στο σημείο 12 θα ήθελε μάλλον το σημείο 12 να μεταφερθεί αύριο μετά το σημείο 17 μη υπάρχουν σας αντιρρήσεως, θα το κάνουμε αυτό, αν δεν θέλει κανείς να παρεύει. Επομένως, μετά από αυτή την αλλαγή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών βάσει της πάγιας πρακτικής, αν δεν εγερθεί κάποια αντίληση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούνται τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί. Έρχομαι στο σημείο 3, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας πω πρώτο, πρώτα ότι και η τρέχουσα συνεδρίαση βρίσκεται στο διαδίκτυο, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και ιδίω επειδή έχουμε τη συζήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Καναδά, την ΣΕΤΑ, θα έχουμε περισσότερη τηλεθέαση από ό,τι έχουμε κανονικά. Και γι' αυτό σας καλωσορίζω όλους που μας παρακολουθείτε από το Λονδίνο ως τη Λισαβόνα, αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίασή μας. Και με με ανάμεικτα συναισθήματα πρέπει να σας πω το εξής. Η Τατιάνα Ματσίκοβα, η οποία τόσο πολύ καιρό ήταν μέλος της γραμματείας μας και μας υποστήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δυστυχώς έχει φύγει από τη γραμματεία μας και είναι τώρα επικεφαλής μονάδος στην μονάδα διεύρυνσης της Γενικής Διεύθυνσης expo Ευχαριστούμε πολύ Τατιάνα λοιπόν για το έργο σου και κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σου καθήκοντα. eine inhaltliche... Μία ακόμα ανακοίνωση. Στον ΠΟΕ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για τα αγαθά του περιβάλλοντος. Έχουν υπάρξει σημαντικές πρόοδοι σε αυτές πρόοδη στις, ε, στις ε, συζητήσεις στη Γενέβη. Υπήρξε μια νέα πρόταση από τις 29 Σεπτεμβρίου. Το κείμενο αυτό τώρα είναι υπό επεξεργασία και ελπίζουμε ότι στις 20 Οκτωβρίου θα έχει πάρει την τελική της μορφή. Επομένως, αυτή η συμφωνία βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σημείο 4 τώρα. Διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριλόγου. Έχουμε μία μονάχα τέτοια συζήτηση που συνεχίζεται σε επίπεδο τριλόγου και δεν έχει ακόμα περατωθεί. Η ομάδα διαπραγμάτευσης μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε μια κοινή πολιτική δήλωση στις 15 Ιουνίου για τα λεγόμενα ορυκτά από χώρους συγκρούσεων Έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες λοιπόν και στις 27 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα μια τεχνική συνεδρίαση όπου συζητήσαμε τα ουσιαστικά σημεία και τα έχουμε εδραιώσει στο κείμενο και σήμερα μετά από τη συνεδρίασή μας οι συγητές, ο εισηγητής και οι οι εισηγητές θα συναντηθούν και θα εξετάσουν τις πρόοδους στην εργασία για το θέμα αυτό. Θα την αξιολογήσουμε την πρόοδο Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγγνώμη, προβλέπεται η επόμενη τέτοια συνάντηση, ώστε ελπίζουμε ότι τον Νοέμβριο ενδεχομένω θα είμαστε σε θέση να οριστικοποιήσουμε και το νομοθετικό κείμενο και αυτό θα είναι ένα θετικό βήμα για να εξασφαλίσουμε μια πολιτική δικαίου εμπορίου για τις πρώτες ύλες που προέρχονται από περιοχές σειράξεων. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 5, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κέντρο βάρους της σημερινή μας ε, συνεδρίασης. Πρόκειται για τη συζήτηση ή για μια περαιτέρω συζήτηση σε σχέση με την επικείμενη Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, γνωστή ως ΣΥΤΑ. και η οποία ε, βρίσκεται ενώπιόν μας και επίκειται η απόφαση του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία αυτή. Όπως ξέρετε, από το 2009 έχει ξεκινήσει η συζήτηση με τον Καναδά για μια συνολική συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα. Ένα προσωρινό κείμενο δημοσιεύτηκε το 2014 και χάρη στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρασε το κείμενο αυτό μια, ένα νομικό έλεγχο, ο οποίος οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές για το κείμενο αυτό. Οι διαιτητές για το σύστημα επίλυσης διαφορών έχουν αφαιρεθεί από το κείμενο και υπάρχει μια νέα πρόνοια για τακτικούς δικαστές οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο αυτό. Από τις 22 Φεβρουαρίου λοιπόν υπάρχει το τελικό κείμενο το οποίο από τον Ιούλιο είναι διαθέσιμο και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου έχει ακολουθήσει μια σειρά συζητήσεων, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο βέβαια, αλλά και μεταξύ των φορέων της κοινή γνώμης. Η τωρινή κατάσταση τώρα είναι ότι στο Συμβούλιο οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν προχωρήσει για την απόφαση του Συμβουλίου στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 12 Οκτωβρίου συναντιέται η Κορεπέρ, η οποία κανονικά θέτει το γενικό πλαίσιο για την απόφαση του Συμβουλίου που θα λάβει χώρα, όπως είπα, στις 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο είναι έτοιμο να υπογράψει αυτή τη συμφωνία και αν τα 28 κράτη-μέλη Τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα θελήσουν να προσυπογράψουν αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες για την φύση αυτής της ε, συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία θεωρείται μεικτή συμφωνία. Υπάρχει λοιπόν και ένα τμήμα Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα όπου υπησερχόμεθα και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τι ελεκτικέ μα εξουσίε και τη δυνατότητα συναπόφαση, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία υπόκεινται στην εθνική δικαιοδοσία και ω εκ τούτου Πρόκειται για μια συμφωνία μεικτού χαρακτήρα και γι' αυτό απαιτείται και η ομόφωνη ε, συμφωνία όλων των κρατών μέλων. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που θέλω να σας υπενθυμίσω. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα το οποίο υπόκειται στην ευρωπαϊκή ευθύνη, την ευθύνη των ευρωπαϊκών φορέων και ένα μικρότερο τμήμα το οποίο έχει να κάνει με την εθνική ευθύνη Επομένως, η Επιτροπή μας θα πρέπει να λάβει υπόψη ποια τμήματα της συμφωνίας εμπλέκουν την εθνική αρμοδιότητα και ποια είναι αυτά τα οποία εμπλέκουν την ενωσιακή αρμοδιότητα. Στις 18 Οκτωβρίου θα αποφασίσει το Συμβούλιο για τα θέματα τα οποία είναι εθνικής αρμοδιότητας και στη συνέχεια το μεγαλύτερο τμήμα εμπλέκεται στην ενωσιακή αρμοδιότητα, οπότε μετά από την ε, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να εφαρμοστούν και αυτά τα τμήματα. Και επίσης θέλω να σας πω δεν θα υπάρξει προσωρινή εφαρμογή οποιασδήποτε πρόνοιας του, ε, της, του σχεδίου συμφωνίας μέχρι όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει θετικά. Αυτό είναι απόρρια της ε, Συνδίκης Λισαβόνας από το 2009 και εμείς θα πρέπει να λάβουμε την απόφαση για οποιαδήποτε προσωρινή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Σε εθνικό επίπεδο μπορεί να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή εξάλλου μόνο όταν γίνει επιτυχώς η κύρωση από τα κοινοβούλια των 28 κρατών μελών. Τρίτο στοιχείο. Οι υπουργοί που θα λάβουν μέρος στην συνολική απόφαση <clears throat> θα εκδώσουν και μία ανακοίνωση, μία δήλωση στις 18 Οκτωβρίου που θα παρουσιάζει και την συμφωνία αυτή προς την κοινή γνώμη. Αν υπάρξει λοιπόν μία συμφωνία επί, επί του θέματος αυτού, <clears throat> θα ακολουθήσει και η υπογραφή στις 27 Σεπτεμβρίου, σε Οκτωβρίου σε επίσημη τελετή και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει την εξέταση του συνολικού πακέτου της ε, συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση για ορισμένα τμήματα αυτής της συμφωνίας για να προετοιμάσουμε και τις ε, ε, επερχόμενες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι και για το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας πέντε εμπειρογνώμονες ο κύριος Πέσονεν, ο οποίος είναι γενικός γραμμα της ε, ΚΟΠΑ, ΚΟΠΑ Κογκέκα, της Αγροτικής αυτής Ένωσης, που είστε. Εδώ. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Λουίζα Σάντος, η Διευθύντρια για Διεθνή Θέματα της Business Europe. Καλώς ήλθατε. Ο κύριος Ιαν Πρίτσορτ, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Πένι Κλάρκ, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την παροχή, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και η, κυρία Νίνα Ρένσο από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την υγειονομική περίθαλψη η οποία δεν έχει έρθει ακόμα αλλά περιμένω ότι θα εμφανιστεί όσο να Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες καταρχήν για πέντε λεπτά ο καθένας. Μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάμπρεξ, ο οποίος είναι ο μας και στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων και πάλι θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε τρία λεπτά και μετά αν θέλουν μεμονωμένοι βουλευτές και αυτοί μπορούν να λάβουν το λόγο για να θέσουν τις παρατηρήσεις τους. <clears throat> Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος ε, πρεσβευτής του Καναδά είναι μαζί μας. Καλώς ήλθατε. Και μετά από την συζήτησή μας θα του δώσω και του πρεσβευτή του Καναδά τον λόγο, όπως επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλος θα επανέλθουμε στον εισηγητή μας. Αυτή λοιπόν είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ε, εμπλεκομένων στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και ξεκινάμε με τον κύριο Πέσονεν, ο οποίος έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Dear Chairman, members of the European Parliament, it's indeed a pleasure. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα το πρωί και μπορώ να σας μιλήσω για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ εμείς η ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ που είναι η Ένωση των Συνεταιρισμών Αγροτών και των ε, Ενώσεων Συνεταιριστικών Αγροτικών Επιχειρήσεων θεωρεί ότι αυτό το θέμα είναι στρατηγικής σημασίας. Πριν ασχοληθώ με τα συμπεράσματα θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία στοιχεία τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Ε, μπορεί να γνωρίζετε ότι εν γέννη οι γεωργικές κοινότητες ενδιαφέρονται για την πρόσβαση στην αγορά. Το της συμφωνίας που αφορά σε αυτό το κομμάτι και είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι αν θέλετε. Ειδικά σε ό,τι αφορά το βόλιο και το χοιρινό κρέας, θεωρώ ότι, αυτά τα τμήματα της συμφωνίας μπορεί να πλήξουν την ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι οι Καναδοί διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει πάνω σε κάποια από τα πρότυπα που τα θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά στην Ευρώπη, ειδικότερα όσον αφορά στο βόλιο κρέας χωρίς ορμόνες, και στη σωστή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων ε, για να περιορίζεται ο όγκος των εισαγωγών στην εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες ανησυχίες για τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής, υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει το βόλιο κρέας ελεύθερο ορμονών και η σχετική απαγόρευση και το πώς οι Καναδοί ομόλογοι μας έχουν δεχθεί αυτή την αρχή το ίδιο ισχύει και για το χοιρινό κρέας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αγορά, τους ευρωπαίους καταναλωτές και πόσο μπορεί να διαταραχθεί αυτή. Θέλουμε να σας υπογραμμίσουμε αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι Καναδοί ε, διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει τουλάχιστον εν μέρη να είναι ενιαία οντότητα, να θεωρείται ως ενιαία οντότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε εξαγωγέ σε τρίτε χώρε. Θεωρούμε ότι είναι καθοριστική σημασία σε αυτό το σκέλο, αυτή η διάσταση και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στι συζητήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική τη πολιτική. Ω προ τα γαλακτοκομικά, τα συμφέροντά μα είναι κάπω πιο επιθετικά. Και υπό αυτή την έννοια καλωσορίζουμε τη βελτιωμένη πρόσβαση στην καναδική αγορά. Ε, ορισμένα έχουν πλήρη, πλήρως απελευθερωθεί και χαιρόμαστε γι' αυτό στο Καναδά και ε, ειδικά για το θέμα των τυριών, τυριά πάντως, ε, παντός είδους, χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί μπορούμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά τη διαχείριση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων για να δει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις επιταγές για το βόλιο και χοιρινό κρέας. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση στην καναδική αγορά βλέπουμε την πλήρη απελευθέρωση του αμπελοϊνικού τομέα και αυτό είναι σημαντικό διότι πριν από λίγα χρόνια μετά από την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ίνος υπέφερε ιδιαίτερος από τις απαντήσεις και τις αντιδράσεις ε, των Καναδών. Και από αυτή την ενέα χαιρόμαστε, διότι υπάρχει μια πιο σταθεροποιημένη προσέγγιση, ε, μια πιο σταθεροποιημένη ε, ε, αγορά, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην καναδική αγορά, έχουμε state level 2 στις περισσότερες περιφέρειες. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό και για άλλες εμπορικές ε, συμφωνίες πάνω στις οποίες εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Είναι μεγάλες οι βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες χαίρονται διότι υπάρχει πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ε, ε, λιπασμάτων και έχουμε upstreaming στη βιομηχανία. Να καταλήξω λέγοντας ότι από γεωργική σκοπιά είναι μια συμφωνία πακέτο η ΣΥΤΑ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Κάποια δύσκολα σημεία παραμένουν ως προς την πρόσβαση στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ακρατάντως ότι έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ως αξιόπιστος εταίρος σε διεθνές επίπεδο ακριβώς το πεδίο που υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κομίζει τα μεγαλύτερα ωφέλη στην οικονομία μας. Δηλαδή εξαγωγές υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών προϊόντων που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα σε τρίτες χώρες και τρίτες αγορές. Ο Καναδάς θεωρούμε ότι θα διευκολύνει ε, τον προσανατολισμό μας στις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες στις υπόλοιπε πολιτικός σημαντικός εταίρος, ε, ίσως λιγότερο ευαίσθητα τα ζητήματα που μας συνδέουν με τον Καναδά από ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με άλλους εταίρους. Mm. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε τη ΣΕΤΑ δεδομένων των διοικητικών ε, διαδικασιών που θα πρέπει να διευκρινιστούν και να τύχουν απολύτου παρακολούθησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάντους έχει το λόγο τώρα. Καλημέρα σε όλους. Ε, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Θα έχετε λάβει την κοινή δήλωση των ευρωπαϊκών και καναδικών επιχειρήσεων μεγάλων και μικρών το οποίο αποτυπώνει και τη στήριξη που δίνουν και οι δύο κοινότητες στην συμφωνία αλλά θα ήθελα να εξηγήσω σύντομα γιατί υποστηρίζουμε τη συμφωνία αυτή και θα δώσω δύο παραδείγματα όταν πριν από 7 χρόνια ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις, ε, υπήρχαν μεγάλες επιφυλάξεις ε, και από τις δύο πλευρές κατά πόσον θα μπορούσε ο Καναδάς ιδιαίτερα περιφερειακά και ιδιαίτερα στις δημόσιες προμήθειες και τις υπηρεσίες. Όμως ο Καναδάς κατάφερε να καλύψει αυτές τις, τα πεδία της περιοχή το οποίο μας επέτρεψε να έχουμε εξαιρετική πρόσβαση στην αγορά σε πεδίο που είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και που συνήθως ε, είμαστε συλλογικά επιθετικοί. Δημόσιες προμήθειες λοιπόν, ένα πεδίο κλειδί στο οποίο επιτύχαμε αυτά που επιδιώξαμε. Για τις υπηρεσίες δεν θα πάω σε λεπτομέρειες. Για την επαγγελματική αναγνώριση, ε, οι συνάδελφοι στο πάνελ προφανώς θα μας φούν περισσότερα, αλλά είναι και αυτή μια περιοχή στην οποία έχουμε πολλά επιθετικά συμφέροντα. Κάποιες φορές δεν υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες, στις ε, παροχές υπηρεσιών σε κάποιες χώρες. Νομίζω ότι και εδώ θα επιτύχουμε περισσότερη διαφάνεια για τους παρόχους, αλλά το εξής στοιχείο θα υπογραμμίσω η προσωρινή απόσπαση είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν ξεκινούν εκτός των τυχών γιατί γνωρίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε εμπειρογνωμοσύνη know-how. Και εδώ είναι ένα πολύ καλό στοιχείο συγκριτικής αξιολόγησης για τις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε και στις ονομασίες προέλευσης και εγώ καθότι είμαι Πορτογαλίδα και είμαι από τον Νότο, τον Ευρωπαϊκό, είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο επίσης επιτύχαμε μια σειρά από σημαντικά σημεία, αλλά 173 παρότι δεν τις καταφέραμε όλες, ενδείξεις είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και είναι και προηγούμενο για άλλες συμφωνίες για το Πόρτο, για την Γκράνα Παντάνο, για το ελαιόλεδο... για την Σαπάνια, για μια σειρά προϊόντα στα οποία έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιθετικό συμφέρον. Αυτό το αναγνωρίζει και ο Καναδάς και είναι σημαντικό. Πάω τώρα στους δασμούς. Και μιλώ για ένα τομέα που πάνω απ' όλα αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κλωστοϊφαντουργία, αν μιλούμε για την εξαγωγή ενός ε, φιλανδικού προϊόντος, για παράδειγμα, στον Καναδά, μεταξύ του 18 και του 70% δασμούς πρέπει να καταβάλουμε στον Καναδά. Σε αντίθεση με τον Καναδά. Ή η συμφωνία μας επιτρέπει duty free εξαγωγή. Και είναι ένα ισότιμο παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές και τις καναδικές επιχειρήσεις. Και ρυθμιστικά επιτύχαμε βελτιώσεις και θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερες τιμές για τα προϊόντα μας. Για τα είναι για παράδειγμα. Νωρίτερα, όταν θέλαμε να εξαγάγουμε, είχαμε δεσμευτικά την παρτίδα του προϊόντος, την αποστολή, να τη μοιράσουμε μεταξύ προϊόντος εξαγωγής και τοπικών Τώρα δεν έχουμε αυτή τη δέσμευση και επομένως είναι ακόμη πιο ισότιμο το παιχνίδι μεταξύ των ευρωπαϊκών και καναδικών επιχειρήσεων και πάλι. Αυτή λοιπόν η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία, η ΣΕΤΑ για να συνεννοούμεθα, μας διευκολύνει σε διάφορες περιοχές και σε διάφορα σημεία και προσπαθούμε και από τις δύο πλευρές να καλύψουμε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στην κοινή γνώμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, για την προστασία των επενδύσεων, για μια σειρά από θέματα. Και νομίζω ότι και στη διακήρυξη και στο περιεχόμενο της συμφωνίας αμφότερες πλευρές έκαναν ό,τι μπορούσαν και κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν τις ανησυχίες αυτές. Πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη, πολύ προοδευτική συμφωνία που επιτυγχάνει αυτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και των δύο πλευρών και νομίζω και για την κοινωνία συνολικά. Ευχαριστώ κύριε Σάντος. Ο κύριος Πρίτσαρντ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης όπου τα μέλη μας είναι από τεχνικά επιμελητήρια, από δημόσιες αρχές και ανεξάρτητες επαγγελματικές οργανώσεις επίσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδίω στην ΣΥΤΑ είναι η επαγγελματικού χαρακτήρα υπηρεσίες και είμαστε υποδια... έχουμε υποδιαπραγμάτευση μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με τους ομολόγους μου του Καναδά την ε, υπηρεσία αδειοδότησης αρχιτεκτών στο Καναδά. Ο, το κύριο μέλημά μας είναι συνέχεια των προσπαθειών που έχουμε κάνει μετά από το 1990 όταν θελήσαμε να αναπτύξουμε διεθνή πρότυπα μέσω της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων και της Χάρτας Παιδείας της ε, UNESCO. Η βάση για τη συμφωνία μας είναι χρησιμοποίησαμε ένα κοινό έντυπο το οποίο υποβλήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου από τις ε, οργανώσεις μας και είναι το παράδειγμα XY στο κεφάλαιο για τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Προβλέπει πέντε χρόνια επαγγελματικής εκπαίδευσης και δύο χρόνια μαθητεία μετά από αυτό. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τώρα είναι κυρίως αποτελέσματα των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα. Τα... Φυσικά τα συστήματα αυτά είναι αρκετά ομοιογενείς στις επαρχίες του Καναδά και τι πολιτείε του Καναδά, ενώ στην Ευρώπη υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας, επομένως έχουμε τελείω διαφορετικέ προσεγγίσει στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων και στι ρυθμίσει. Πολλέ χώρε έχουν μία εκ των προτέρων ρύθμιση επί τη βάση των ακαδημαϊκών τίτλων, άλλε εκ των υστέρων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του επαγγελματό. Και μερικά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μία σαφή έννοια μαθητία ή αδειοδότηση για του αρχιτέκτονε. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και αυτό παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι τα, πλαίσια, τα πρότυπά μας είναι πολύ ψηλά και τα συστήματά μας παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εναρμοστεί είναι αντίστοιχα αυτών του Καναδά. Έχουμε καταφέρει να γίνει, δεκτή, να γίνει δεκτό το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα στο σημείο 46 αναφέρει ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων και επίσης σε ό,τι αφορά την ερεσιμότητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν, ε, έχουν διπλώματα και αυτοί που έχουν δικαιώματα βάσει του άρθρου 6 θα είναι επιλέξιμοι για την αναγνώριση. Κάτι ακόμα που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα περιχαρακώσουμε την ειδική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς. Παραγματικά χάρη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση συμβολέων, τα ε, έγγραφα, του, τα αρχιτεκτονικά έγγραφα και σχέδια. Αντί να έχουμε λοιπόν διαδικασία προσωπικού ελέγχου μέσω συνεντεύξεων, αποφασίσαμε να έχουμε ένα σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να γίνει μια <clears throat> εκπαίδευση, μια σύντομη εκπαίδευση επιγραμμικά στο διαδίκτυο δηλαδή για τους αρχιτέκτονες. Και επίσης έχω ήδη ενημερώσει την ομάδα των συντονιστών για το γεγονός ότι το, η υπηρεσία διοδότησης του Καναδά θα συναντηθεί στο τέλος του μήνα για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Θα πληροφορήσει και τις αρμόδιες αρχές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ένωση Εκτεκτώνων θα ελπίζει να μπορέσει να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία το Δεκέμβριο και επίσης στην ΟΤΑΒΑ την επόμενη χρονιά θα γίνει δεκτή αυτή η απόφαση και από την καναδική πλευρά. Το τελευταίο θέμα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί είναι πώς θα γίνει η εφαρμογή επί τη βάση του διεθνούς δικαίου αυτής της συμφωνίας. Εμείς θέλαμε να αναφέρουμε Στι Ομοσπονδιακέ αρχέ του Καναδά και στην Κομισιόν τη σύμφωνη αυτή για να παραπευθεί στην αρμόδια Επιτροπή MRA που έχει δημιουργηθεί βάσει τη ε, ΣΥΤΑ. Παρ' όλα αυτά όμω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη <clears throat> το γεγονό ότι τα επαγγελματικά διπλώματα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτιών και των πολιτιακών οργάνων αδειοδότησης στον Καναδά. Μπορεί λοιπόν να θελήσουν να κάνουν μια άμεση συμφωνία με εμά και να δημιουργήσουν τη δική τους ε, Επιτροπή Διακυβέρνησης για την, τον εποπτεία αυτής της συμφωνίας. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουν και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριληφθούν σε αυτή τη συμφωνία μέσω της Επιτροπής της ε, ΣΥΤΑ για τα θέματα αυτά. Παραμένει αυτό λοιπόν ε, κρέμας και είμαστε σε επαφή με την Trade και διερευνούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να οριστικοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρίτσοτ. Η κυρία Κλόκ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, για την συμμετοχή σημερινή συζήτηση. Έχω κάποιες διαφάνειες και ένα έγγραφο που εξηγεί κάπως τα σημεία. Η Τζοάννα θα έχει την ευγενή καλοσύνη να με βοηθήσει με τις διαφάνειες. Λοιπόν, ο δικός μας φορέας, όπως και αρκετέ άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν είναι υπέρ τη συμφωνία αυτή. Σα συστήνουμε να μην την στηρίξετε. Έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό ώστε να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτό και να επηρεάσουμε την πορεία της διαπραγματεύσης, της συζήτησης και να συνοψίσουμε, <clears throat> να συνοψίσουμε πολύ σύντομα Δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ εκπροσωπώ τους εργαζομένους σε πάρα πολλές δημόσιες, τοπικές, περιφερειακές αρχές, ύδατο, ε, υγειονομικέ, Έχουμε συνεργαστεί και με άλλα συνδεκάτα στην παιδεία, στις μεταφορές. Έχουμε μεγάλη ανησυχία για την ικανότητα νομοθέτησης, ρύθμιση στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και κυρίω στου ιδιωτικού παρόχους δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό μαζί με τον αρνητικό κατάλογο και τις ε, standstill ρήτρες που φαίνεται η Κομισιόν να αρέσκεται πολύ, να τις πολλαπλασιάζει, είναι πολύ προβληματικές. Και αν δούμε και τον φορέα, το δικαστήριο των επενδυτών, ε, αυτό υπογραμμίζει την όλη ανησυχία αυτή. Η τρίτη δέσμη ανησυχίας είναι η ελλειπής προστασία για τους ε, εργαζομένους και για το περιβάλλον. Αυτές τις ανισχύες τις μοιράζεται μια ευρύτατη, ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικό και είχαμε και μια κοινή δήλωση με την Ένωση Καταναλωτών φορείς του περιβάλλοντος, είμαστε μέλη της ε, ΤΟΥΚ ε, και άλλων ομοσπονδιών πάρα πολλές ενώσεις, πάρα πολλοί φορείς ε, μοιράζονται τις ανησυχίες αυτές και μάλιστα και από την πλευρά των Καναδών. Έχουμε δουλέψει από το 2008 με Καναδικές Ενώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημείο που αναφέρθηκε από τους ομιλητές προηγουμένως. Έχουμε πάει σε αυτή την κατεύθυνση επιθετικών και αμυντικών συμφερόντων. Εμείς θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι και οι πολίτες έχουν συμφέροντα κοινά σε διάφορες χώρες. Και έχουμε προτείνει στους Καναδούς ομολόγους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το δίκαιο εμπόριο, για το ισότιμο εμπόριο, να έχουμε μια κοινή στάση. Στα πλαίσια της συμφωνίας όλα αυτά δεν έχουν μετατραπεί, αν θέλετε, μεταφραστεί στην προστασία των κοινών κοινωνικών συμφερόντων με ισορροπημένο τρόπο. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, αλλά καθότι έχουμε αυτήν τη δήλωση, αυτή τη φάση τώρα, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει κανείς την ψυχραιμία του και να αξιολογήσει την όποια δήλωση, έχοντας υπόψη το, το, το, περιεχόμενο του κειμένου και προσπαθώντας να απαντήσει επί τα θέματα, τα προβλήματα που υπήρχαν το κείμενο και αν όχι πρέπει κανείς να εξαγάγει τα συμπεράσματά του. Επομένως, εγώ συνέλεξα κάποια στοιχεία και θα τα βρείτε στο έγγραφο που έχουμε μοιράσει από τη συμφωνία, διότι υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια στοιχεία αμφιλεγόμενα, ιδιαίτερα σχετικά με τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη δηλωσία. Και θα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το νερό ή όλες οι εκστρατείες για το δικαίωμα στην υδροδότηση και ε, ε, που θα έπρεπε να αποκλειστεί κανονικά από τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά αυτό δεν είναι έτσι. Αν δείτε τη ΣΥΤΑ, λέει ότι εάν το νερό είναι ανοιχτό στις εμπορικές χρήσεις, θα πρέπει να ισχύουν οι ρήτρε της συμφωνίας. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα στην Δανία και στην Ουγγαρία, για τη συμφωνία που έχουμε για τα υγειονομικά συστήματα, για την κοινωνική προστασία, όπου ζητείται δηλαδή μακροπρόθεσμα από τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστεί το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας με, με τα πλαίσια συμφωνιών σαν και αυτήν. Και για να ολοκληρώσω, Τζοάννα, α, ευχαριστώ επανέρχομαι στις δημόσιες υπηρεσίες για να πω ότι υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό. Του κεφαλαίου 17 της συμφωνίας επί της ανταγωνιστικότητας, αριστερά, που βασίζεται στους κανόνες για τις ε, κρατικές ενισχύσεις, που δίνει κάποιες, κάποιους περιορισμούς σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει το θέμα των δημοσίων υπηρεσιών ενώ δεξιά στη στήλη βλέπετε μια πιο δημοκρατική θα έλεγα ερμηνεία των δημοσίων υπηρεσιών που λέει ότι οι πολίτες εφασίζουν, δημοκρατικά φυσικά, τίποτα δεν μπορεί να επιβληθεί και αυτό είναι το διακύβευμα στα πλαίσια τη συμφωνία αυτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κλάρκ, η κυρία Ρέντσαρτ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Με λένε Λίνα Ρέντσοντ. Είμαι Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Δημόσιας Υγείας 90 οργανώσεις που εκπροσωπούν τις επαγγελματικές, τους επαγγελματικούς συλλόγους των ιατρών, νοσηλευτών, ειδικών επαγγελματιών της υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή και παρέχουν φροντίδα και υπηρεσίες υγείας στις πιο ευπαθείς ομάδες. Εκπροσωπούμε ενώσεις ε, εξειδικευμένες σε συγκεκριμένες νόσους και μας ενδιαφέρει η καλή ποιότητα ε, των υπηρεσιών υγεία, έτσι ώστε όλοι στην Ευρώπη να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία. Δεν είμαστε κατά του ελεύθερου εμπορίου, το λέω ευθύ εξ αρχή. Θα θέλαμε όμως να δούμε τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις να είναι έτσι ώστε να είναι ευεργετικέ για τη δημόσια υγεία και να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Και δεν πιστεύουμε ότι το κείμενο της ΣΥΤΑ, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή, επιτυχάνει αυτή την ισορροπία. Ακόμα και μετά τις τελευταίες ερμηνείες που έχουν δοθεί, δεν έχει δικλείδες ασφαλείας απαραίτητες για να προστατευτεί και να βελτιωθεί η δημόσια υγεία. Δεν είναι μια καλή συμφωνία υπ' αυτή την έννοια. Δεν θα μιλήσω λεπτομεριακά για τις υπηρεσίες, το είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, όμως συμφωνούμε με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και κυρίως με τα υπόλοιπα. Προστασία των επενδύσεων. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να ζητούν αποζημίωση για μέτρα δημόσιας πολιτικής, μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας όταν οι επενδυτικές τους προσδοκίες διαψεύδονται. Δεν είναι απαραίτητο ε, κάτι τέτοιο μέσα σε μια εμπορική συμφωνία όριμων οικονομιών που είναι κράτη δικαίου και έχουν όριμα δικαστικά συστήματα. Δεν χρειάζεται μια τέτοια ρήτρα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει ένα συγχώριος μηχανισμός και ε, εκ των προτέρων συμμετοχή του δικαστηρίου ε, του Ευρωπαϊκού έτσι ώστε μετέπειτα και μεταγενέστερα δικαστήρια να ερμηνεύουν σωστά την ευρωπαϊκή νομολογία. Ε, μπορεί να είναι θετικός ο, θετικός ο αντίκτυπος στις τιμές του καταναλωτή. Υπάρχουν όμως δύο εξαιρέσεις που αξίζει να εξετάσουμε. Πρώτον, φάρμακα και ιατρικές συσκευές Υπάρχουν ευαίσθητες διατάξεις για την εθελούσια συνεργασία. Αυτό είναι κάτι που ήδη συμβαίνει και εκτός ε, εμπορικής συμφωνίας με Καναδά και θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ανεξαρτήτως του, της έκβασης. Άλλωστε παραμένει η ανησυχία της πρόσβασης στα φάρμακα. Η δαπάνη φαρμακευτική στον Καναδά, η κατακεφαλή η δεύτερη υψηλότερη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Προβλέπονται αυξήσεις κατά 6-13% των φαρμάκων στο Καναδά. Θα θέλαμε να γίνει σχετική μελέτη και για το τι ε, θα συμβεί στην Ευρώπη. Γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία τελικά θα κάνει τις τιμές των φαρμάκων να εκτοξευθούν και να μην μειωθούν. Σίγουρα το αυξημένο εμπόριο και η αυξημένη προσβασιμότητα θα είναι ε, ε, εις βάρος της δημόσιας υγείας. Αναφέρομαι κυρίως στα προϊόντα καπνού, αλκοόλ και προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η άρση των δασμών θα έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία. Δεν λέμε να αυξηθούν οι δασμοί ή να διατηρηθούν, ωστόσο είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι θα έχει αντίκτυπο στη δημόσια υγεία να έχει κανείς ώστε να τον μεγαλύτερη και φτηνότερη πρόσβαση σε προϊόντα διατροφικά σε, με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, σε προϊόντα καπνού ή σε προϊόντα αλκοόλ. Όλα αυτά θα πλήξουν τη δημόσια υγεία. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και θα έχουν στη συνέχεια, ε, θα υπάρχουν φαινόμενα αύξησης των εθισμών, του καρκίνου, του διαβήτη, ε, διαφόρων νοσημάτων που ούτως ή άλλως επιβαρύνουν τα εθνικά συστήματα υγείας και μπορούν να απειλήσουν την ύπαρξή τους αυτή καθεαυτή λόγω του μεγάλου βάρους τους στο, ε, στη δημόσια υγεία. Θα πρέπει ε, λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση να ρυθμίζει για να αντισταθμίζει αυτές τις απώλειες και αυτό τον αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Εάν ε, πάρουμε μέτρα ε, για να υπάρχει αναγραφή της επικοινωνία στα προϊόντα καπνού, εάν πάρουμε μέτρα για να υπάρχει μια συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή στην πώληση αλκοόλ, προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, θεωρούμε ότι μετά θα, οι επιχειρήσεις θα ε, αμφισβητήσουν αυτού του είδους τα μέτρα και θα πάμε στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών ως χώρες, κάτι το οποίο θα αποτελέσει μεγάλο χτύπημα στη δημόσια υγεία, μεγάλο πλήγμα. Σε κάθε περίπτωση ε, ε, μπορεί να είναι θετικά αυτά για την Ευρωπαϊκή Γεωργία τα περιεχόμενα, για το βόηο κρέας και ούτω καθεξής, αλλά δεν ρυθμίζεται το πρόβλημα της πολύ ισχυρής αντίστασης στα αντιβιωτικά, λόγω της ευρείας και αλόγης της χρήσης τους. Θεωρούμε ότι η ερμηνευτική δήλωση είναι καθοδηγητική αλλά όχι καθησυχαστική. Υποτίθεται ότι πρέπει να καθυσυχάσει εμάς που θέλουμε το, να διατηρηθεί το δικαίωμα της νομοθετικής ρύθμισης για την ε, πολιτεία, την εκάστοτε. Σε κάθε περίπτωση δεν επαρκούν αυτά, δεν είναι αρκετά σαφές το κείμενο δεν νομίζουμε ότι αυτή η ερμηνευτική δήλωση έχει νομικό βάρος, νομική δεσμευτική ισχύ. Καλούμε λοιπόν τα μέλη να ζητήσουν νομική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας όλες αυτές τις ανησυχίες των καταναλωτικών οργανώσεων που πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η συμφωνία. Ευχαριστώ λοιπόν. Έχουμε ακούσει τους πέντε πυρογνώμονες. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή, μετά στους σκιώδεις από τις πολιτικές ομάδες. Τρία λεπτά παρακαλώ. Εάν έχετε να θέσετε ερωτήματα, παρακαλώ διατυπώστε τα μεσαφήνια και πείτε προς ποιον απευθύνεται το ερώτημα αυτό. Μην θέτετε ερωτήματα συλλήδιν προς όλους. Αλλά πείτε σε ποιο, ποιος θέλει να σας το απαντήσει και φυσικά μπορούμε να ζητήσουμε και από την Κομισιόν και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος διαπραγματευτής της Κομισιόν οπότε η Κομισιόν είναι και αυτή σε θέση να απαντήσει ελπίζω σε ερωτήματα Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Πάμπλεξ, στον εισηγητή μας σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση σήμερα το πρωί, γιατί μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες της ε, συμφωνίας δημόσια τα τελευταία δύο χρόνια μετά από την δημοσίευση του κειμένου μπορούν έτσι να, να διευκρινιστούν καλύτερα οι θέσεις μας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους ομιλητές οι οποίοι έλαβαν το λόγο και μας είπαν, μας δώσαν σημαντικές διευκρινήσεις για αυτήν την σημαντική συμφωνία. Από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σταθώ σε μερικά για μένα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω και βασίζομαι βέβαια σε αυτή την πίστη σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία ότι αυτή η εμπορική συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από οποια οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία. Δεύτερον, αυτή η εμπορική συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ανεπτυγμένων οντοτήτων Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο ανεπτυγμένων εμπορικών οντοτήτων, με ποιον άλλο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι και γεωπολιτικά και οικονομικά είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ ψηλότερα πρότυπα που είναι απαραίτητα για οποιοδήποτε παίκτη στο διεθνές εμπορικό στερέωμα. Όπως βλέπουμε από αυτά που είπαν οι εμπλεκόμενοι θέλουμε όλοι να έχουμε καλύτερα πρότυπα στις πολιτικές μας και ιδίως στις εμπορικές μας πολιτικές. Η ΣΥΤΑ δίνει τη δυνατότητα να συνάψουμε μια συμφωνία που βασίζεται σε υψηλότερα επίπεδα και έτσι με αυτόν τον τρόπο να υποχρεώσουμε άλλες χώρες οι οποίες δεν θέλουν τα υψηλότερα πρότυπα να μας ακολουθήσουν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Επίσης, αυτή η εμπορική συμφωνία και όπως δείχνουν και αναλύσεις έγκριτα περιοδικά όπως το Economist, δίνουν την ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι πάνω απ' όλα ε, συμφωνίες που ευνοούν την <clears throat> φτωχότερη πλευρά και όχι, όπως λένε πολλοί, την πλουσιότερη πλευρά. Εάν εμείς σταματήσουμε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μεταξύ περιοχών και χωρών, οι πρώτοι που θα φυγούν είναι οι φτωχοί. Δεύτερον, θέλω να κάνουμε σαφές ότι αν εγκρίνουμε μια συμφωνία όπως η ΣΥΤΑ, δείχνουμε έτσι ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινή στάση μεταξύ του Καναδά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη. Αλλιώς θα είμαστε απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο και θα οδηγηθούμε σε μια αδύρυτη κάμψη. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και η κοινή γνώμη. Κάτι ακόμα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας και σε όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται στα πραγματικά γεγονότα και όχι απλώς τις πεπιθήσεις και τις προκαταλήψεις ότι δεν είναι μια ιδανική συμφωνία, αλλά και εμείς δεν είμαστε ιδανικά άτομα. Δεν είμαστε ιδανικές χώρες. Και είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς άτομα που δεν είναι ιδα... ιδανικά μπορούν να φτάσουν πολύ κοντά στο ιδανικό. Και από αυτή την άποψη δεν βλέπω αυτή τη συμφωνία που ως μια συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξεκινώντας από την παχυσαρκία και φτάνοντας μέχρι την εκθρόνηση του Ασάτ. Αυτό είναι και η σημασία μια εμπορική συμφωνία, ότι έχει ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να πετύχουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμω μια ανοιχτή πόρτα. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε και να φτάσουμε ακόμα και κοντά στην τελειότητα, ας το κάνουμε. Σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η συμφωνία. Πάντα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης και επειδή υπάρχει αυτή η ευκαιρία βελτίωσης, αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε ήδη τώρα σε μια συμφωνία που δεν είναι ιδανική, αλλά από πολλέ απόψει είναι η καλύτερη δυνατή και πολύ κοντά στην τελειότητα πρέπει να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάμπληξ. για πολύ καιρό υποπτευόμουν ήδη ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ιδανικός χώρος, δεν είναι ο παράδεισος επίγης, λέει ο πρόεδρος. Από τις πολιτικές ομάδες τώρα οι εισηγητές, για τους σοσιαλιστές ο Ντέβιτ Μάρτιν έχει το λόγο τρία λεπτά. Όσο πιο κοντά φτάνει κανείς στην έξοδο, τόσο πιο πολύ μοιάζει με παράδεισο η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ακούσει την άποψη της οργα... των εμπλεκόμενων φορέων και Πιστεύουν οι περισσότεροι ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσβαση στην αγορά είναι καλό για αμφότερα μέρη και για τον Καναδά και για την ΕΕ. Οι δύο τελευταίοι ομιλητέ όμως εξέφρασαν ανησυχίες τις οποίες μοιραζόμαστε και εμείς ως πολιτική ομάδα μας. Ενδιαφέρει το θέμα ε, των διευθετήσεων, των, του δημοσίου τομέα, των δημοσίων υπηρεσιών, Πρέπει να τα μελετήσουμε ε, περισσότερο. Η ερμηνευτική δήλωση πρέπει να είναι δεσμευτική. Εμείς πιστεύουμε ναι. Γιατί πιστεύουν οι ομιλητές ότι δεν είναι δεσμευτική. Και το δικαίωμα του νομοθετεί. Ναι. Το, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει νομοδότηση που θα λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να συνεχίσουν να νομοθετούν όπως πιστεύουν και θα ζητηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές να συνεργαστούν, δεν θα εξαναγκαστούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα δοθεί όθηση στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου τομέα με τη συμφωνία ΣΥΤΑ. Εάν κάποια υπηρεσία επιθυμεί να παραμείνει δημόσια, μπορεί να συνεχίσει φυσικά να το κάνει. και οι ξένοι επενδυτές δεν θα πρέπει να έχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες από τους χώριους επενδυτές. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση των δύο μερών να συνεργαστούν για να υπάρχει κώδικας δεοντολογίας πριν τεθεί σε ισχύ η ίδια η Εμπορική Συμφωνία Καναδά-ΕΕ. Ο Καναδάς έχει ήδη υιοθετήσει τη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε επίπεδο γεωρουσίας ο πρέσβης του Καναδά πρέπει να μας μιλήσει για το πόσο κοντά είναι η χώρα αυτή στην υιοθέτηση ε, της σχετικής σύμβασης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ θετικό το ότι από την εθελούσια βάση περάσαμε σε μια δεσμευτική συμφωνία. Η πολιτική μου ομάδα βεβαίως θα μελετήσει τις ενστάσεις, αλλά σε αυτό το στάδιο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Καναδούς συναδέλφους γιατί ήταν ευέλικτοι και επιθυμούν να ε, συνεχίσουν. Ε, όταν ε, ολοκληρώνεται μια διαπραγμάτευση, συνήθως δεν περιμένει κανείς να δεχθεί το άλλο μέρος να ξανακαθίσει στο τραπέζι. Και ο Καναδάς το δέχθηκε και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Ο κύριος Κέμπερ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μας πλευρά και εμείς χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη συμφωνία αυτή. Ο Καναδάς δεν είναι μια μικρή χώρα, είναι από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια φιλόδοξη συμφωνία, μια φιλελεύθερη συμφωνία και ε, βγάζει από τη μέση 99% των δασμών, 92% των αγροτικών δασμών. Πιστεύω ότι από την άποψη των υπηρεσιών, των ανοίξουν υπηρεσίε δημοσίων προμηθειών, αυτό είναι κάτι επίση πάρα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο. Για μένα λοιπόν είναι μια πολύ καλή συμφωνία, μια υποδειγματική θα έλεγα συμφωνία και γι' αυτό αξίζει της υποστήριξής μας. Πιστεύω ότι και από γενική έποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η TTIP, με την Ινδία να είναι σε τελμάτωση και την Κίνα να μην έχει προχωρήσει καθόλου και την Ιαπωνία να έχει πολύ χαμηλή ανάπτυξη, αν αποτύχει αυτή η συμφωνία της ΣΥΤΑ, τι νόημα έχει να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, δεν έχουμε κανένα ρόλο σε αυτή την αίθουσα τότε, σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την εμπορική συμφωνία. Και τέλος, χωρίς να μπω στο αν είναι παραδείσια ή όχι και για το Brexit που έχει διαφορετική άποψη ο κ. Μάρτιν, η ΣΥΤΑ θα μπορούσε να είναι το υπόβαθρο για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ υποστήριζω μια τέτοια συμφωνία Καναδά συν σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και πάλι ο Καναδάς είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο. Πρέπει να έχει την υποστήριξή μα αυτή τη συμφωνία. Άκουσα, όπω είπαν και οι εμπειρογνώμε, ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε σε συγκεκριμένου τομεί. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank you, um, chairman. Σας ευχαριστώ, η κυρία Στάρκε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω και ακούμε από όλους τους εκπροσώπους ενδιαφερομένων φορέων και είναι και ο ρόλος μας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είμαστε σε επαφή με όλους αυτούς τους φορείς Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη βούληση και την επιθυμία των πολιτών, των επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων φορέων. Νομίζω το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και αποτυπώνει νομίζω και κάποια αποτελέσματα των επιδιώξεών μας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, του αποκλεισμού των δημοσίων υπηρεσιών, Τη προστασία βιωσιμότητα, νομίζω ότι ο κατάλογο είναι μακροσκελή. Τα περισσότερα από τα δύσκολα σημεία, τα κανθόδη σημεία νομίζω ότι έχουν καλυφθεί. Και η προοδευτική κυβέρνηση Τρούντο κάλυψε το χαμένο έδαφος αν θέλετε ή την καθυστέρηση που υπήρχε στην αρχή με πολλές ανησυχίες και νομίζω ότι σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο ανταγωνισμό οικονομικά, αλλά και επί των αξιών και των αρχών μας και των προτύπων. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο εταίρο από τους Καναδούς, ώστε να ενισχύσουμε συνολικά τη διεθνή συνεργασία και να συνεργαστούμε αποκινούμε τους Καναδούς να θέσουμε υψηλότερα πρότυπα για όλους. Έχοντας όμως κατά νου το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας. Επομένως, σκεπτόμενοι τη συμφωνία και τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις όλων μας, νομίζω ότι κάθε ένας από εμά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερψηφίσουμε γρήγορα, γιατί τα ωφέλη είναι εκεί για τους πολίτες μας, οι σχέσεις μας ενδυναμώνονται, ακούμε φυσικά τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες όλων εκείνων που διαφωνούν, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο, εγώ δεν έχω δει ποτέ τέλειο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να υπάρξει ένα απόλυτα τέλειο αποτέλεσμα με τόσο μεγάλο αριθμό φορέων που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή, αλλά και το επικοδομητικό πολιτικό κλίμα και αυτό κάτι αξίζει νομίζω. Και θα έλεγα προς αυτούς που θεωρούσαν ότι μπορούσαμε να επιτύχουμε καλύτερη συμφωνία ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν. Και θα μπορούσαμε προσπαθώντας να κερδίσουμε περισσότερα να διακινδυνεύσουμε τα πάντα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι δηλαδή όταν επικρίνουμε να αναλάβουμε τις ε, ευθύνες του να μην τελικά ολοκληρώσουμε μια τέτοια συμφωνία. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα απειλούσε σημαντικότατα τη δυνατότητά μας να διαπραγματευόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα έθετε το ένα κράτος μέλος κατά του άλλου και τελικά θα κατέτρωγε, θα υπέσχαπτε την ε, ενιαία αγορά, την κοινή αγορά. Και θα μας αποδυνάμωνε από την προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τα πρότυπά μας διεθνώς. Και γι' αυτό πρέπει νομίζω να χαιρετήσουμε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής. Η ε, ε, κυρία, η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Μία ερώτηση θα είχα. Μόνο από του χρόνου θα έχουμε μία απόφαση του δικαστηρίου επί της Σιγκαπούρης. Αυτό τι επιρροή θα μπορούσε να έχει πάνω στην ε, απόφαση αυτή, στην συμφωνία αυτή. Θα μπορούσε να αλλάξει η πορεία μας. Επίσης κάτι φαίνεται να έχει πάει στραβά με τη ΣΥΤΑ. Υπάρχει και αυτή η δήλωση που θα πρέπει να επισυναυθεί στη συμφωνία, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει αυτό το σύστημα διατησίας και τα σχετικά προβλήματα εκεί και η Κομισιόν επίσης αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος, για να μην μιλήσουμε για άλλες πτυχές, θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν. Το αναγνωρίζει αυτό η ίδια η Κομισιόν. Και κατά την άποψή μας ε, έχουμε υποτιμήσει ακόμα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο περιοχές. Θα ακούσουμε όλοι την απόφαση του δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση. Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια πεδία συμφωνία που δεν ε, τα έχουμε εξετάσει καθόλου. Οι διατάξεις racket stand still οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Ε, πρέπει να επιχειρήσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε, να μην ερμηνεύσουμε λανθασμένα, νομικός μιλώντας, το κείμενο αυτό. Τη νομική ισχύ δηλαδή του κειμένου αυτού. Η δήλωση δεν είναι ένα κείμενο νομο, νομοθετικής ισχύω. Ε, είναι μια περιγραφή, μια συνοπτική εικόνα ενός ιδανικού κόσμου θα μπορούσε να πει κανείς. Και μάλιστα θα μπορούσε κανεί να την ερμηνεύσει τελείως αρνητικά. Δηλαδή είναι σαν να δηλώνουμε κάτι χωρίς να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αγνώντας δηλαδή μέσω ποιου πλαισίου διατάξεων θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα το δικαστήριο έχει ήδη πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα επί μιας δήλωσης ε, σαν και αυτήν εδώ. Επομένως, ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μετατρέψει, θα μεταφράσει αυτό το κείμενο, αυτή τη δήλωση σε κάποιον νομικά δεσμευτικά κείμενο και θα επισυναυθεί με κάποιον νομοτεχνικό τρόπο στη συμφωνία. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια λύση και να το κάνει αυτό αποφασιστικά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τη δημοκρατία μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ για τους πράσινους. Για τους πράσινους ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για την ε, συνεισφορά της, τους, τη συζήτηση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο το θέμα της πρόσβασης στην αγορά ακόμα και το αγροτικό λόμπι, αν το μπορώ να το πω έτσι, τονίζει πάντα <clears throat> ότι υπάρχει ένα στοιχείο απαράδεκτο ότι δίδεται η πρόσβαση για το χείριο και το βόλιο κρέας σε μεγάλες ποσότητες από τον Καναδά. Δεν ξέρω αν υποστηρίζετε ακόμα αυτή την ε, θέση, αλλά κάποιοι από τους συναδέλφους σας το έχουν πει. Πολλοί από το γεωργικό τομέα και εργαζόμενοι στο γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Και αυτό θέτει ένα αμφιβόλο θέση απασχόληση μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση επίση σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ γάλακτο η δήλωση των Καναδών ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν ποσοστώσεις γάλακτό. Εμεί. έχουμε τεράστια προβλήματα υπερπαραγωγής γαλακτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στο γαλακτοκομικό τομέα. Και τώρα, αν μα πει ο Καναδάς να σταματήσετε τι ποσοστώσεις, αυτό δεν ξέρω αν θα βοηθήσει την κατάστασή του. Για την παροχή υπηρεσιών και Και εδώ θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα σε αυτή την ερμηνευ... για την ερμηνευτική αυτή δήλωση γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο ελέφαντας που στέκεται με την προβοσκίδα του στην αίθουσά μας. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε, γιατί για πολλούς από τους συναδέλφους μας αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο που θα καθορίσει την θέση τους εναντί της ΣΥΤΑ. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τα σχόλια σας για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υγειονομικές ιδιωσίες υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν πολλές από τις ανησυχίες που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το θέμα. Όταν διάβασα εγώ την ερμηνευτική δήλωση δεν κατάλαβα πως η αίτηση για τις δημόσιες υπηρεσίες συνάδει με το κείμενο, πώς μπορούμε να δούμε στο κείμενο αυτό το οποίο διέρευσε να καλύπτεται αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πώς βλέπετε εσείς αυτή την ερμηνευτική δήλωση και ίσως κάποιος από εσά μπορεί να πει κάτι για το πόσο νομικά δεσμευτική μπορεί να είναι αυτή η ερμηνευτική δήλωση για τη συνεργασία με τον Καναδά. Βεβαίως είμαστε όλοι υπέρ, υποστηρίζουμε, αλλά με τίμημα του να αυξηθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαψης και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι θετικό. Επίσης, για την γεωγραφική προέλευση και την προστασία γεωγραφικής προέλευσης. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός ε, των γεωγραφικών ενδείξεων που θα προστατευτούν. Κάποιες άλλες γεωγραφικέ προελεύσεις, ιδίω από την Ανατολική Ευρώπη, δεν έχουν μπει σε αυτόν τον κατάλογο και είναι αυθαίρετο ο κατάλογο αυτή τη στιγμή. Επίσης για την συνεργασία, όλα αυτά εξαρτώνται από την ύπαρξη ενό καλού διαλόγου με την άλλη πλευρά και γιατί τώρα κάποιο από του συναδέλφου μα που θα πήγαν στη ΣΥΤΑ δεν του δώσαν τη δυνατότητα να μπει στον Καναδά, του ανηθήκανε την είσοδο, αφού έχουμε τον πρεσβευτή του Καναδά, αυτό είναι χρήσιμο. Να μα πει και αυτό στην άποψή του, δεν είναι θετικό και δεν βοηθάει καθόλου να απαγορεύεται η είσοδο στο Καναδά σε ευρωβουλευτέ. Υπάρχει και το θέμα τη αμοιβαιότητα και τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων που εκκρεμεί ακόμα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το, συζητώ, το συζητά αυτό το θέμα, αλλά επειδή έχουμε εδώ τον πρεσβευτή του Καναδά, θα ήθελα και πάλι να έχω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ, λέει ο για την ομάδα του EFDD, η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, πρόεδρε να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους ε, και που περιγράφει και την υφιστάμενη κατάσταση που έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι οπωσδήποτε αυτό το πεδίο της συζήτησης. Αυτό που παρατηρούμε είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών οικονομικών μοντέλων. Και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι μια εισαγωγή αν θέλετε σε μια κατεύθυνση ελευθέρων συναλλαγών ε, το οποίο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλη ανησυχίας περιβαλλοντικής, κοινωνικής ή οποιασδήποτε άλλης. Και εκφράστηκαν φυσικά όλοι οι εκπρόσωποι του κόσμου των επιχειρήσεων πολύ θετικά, ενώ ε, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων και των κοινωνικών φορέων πολύ πιο επικριτικά. Τώρα δεν έχω καμία πρόθεση να ανοίξουμε εδώ μια, ένα κύκλο συζήτησης επί των ελευθέρων συναλλαγών. Το οποίο ε, θα πω απλώς ότι δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι δίνουν τέτοιες συμφωνίες κάποια ε, πλεονεκτήματα στους πιο οικονομικά ευάλωτους, στις πιο ευάλωτες ομάδε τη κοινωνία. Ε, ακριβώς το αντίστροφο φαίνεται να ισχύει από όλε τι ενδείξει που έχουμε στη διαθέσή μας. Όμως, επί τη ΣΕΤΑ θα μπορούσε να μπει κανεί τι είδους οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη επιθυμεί να συνεισφέρει. Μιλούμε για το 0,08 του ΕΕΠ της ε, μεγέθυνσης, της μεγέθυνσης, με συγχωρείτε, ε, που είναι σχεδόν ασήμαντο, σχεδόν αμεληταίο. Επομένω ρωτώ, ρωτώ και του εκπροσώπους των επιχειρήσεων που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, ποια είναι η προβολή ανάπτυξη για τις δικές τους επιχειρήσεις. Γιατί τα συνολικά μεγέθη προβολής είναι σαφή και δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι στοιχεία της ε, Κομισιόν. Και μιλούμε για πάνω από 160.000 επιχειρηματικούς φορείς. Αυτό επί τη βάση μεγεθών, επαναλαμβάνω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χειρότερα στοιχεία από διάφορες ανεξάρτητες ε, εκθέσεις και μελέτες. Επομένως η ερώτησή μου προς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων είναι αυτή. Εσείς τι έχετε προβλέψει, τι έχετε υπολογίσει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα για όλες τις επιχειρήσεις που σήμερα έχουν σταθερή εκπροσώπηση στον Καναδά. Διότι θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές τους, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ποιο είναι ο αντίκτυπο των επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή τη στιγμή παρουσία στον Καναδά. Ενώ μια ερώτηση που θα ήθελα να, να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σχετικά με τη διάταξη reset, αν ακούσαμε καλά, γιατί έχουν ε, ακουστεί διάφορα και θετικά και αρνητικά σχόλια και νομίζω ότι και από των υπηρεσιών είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να διευθυνιστούν απολύτω. E, uh, e Για το ENF, ο κύριο Φέραμο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η συνθήκη της τελευταίας ευκαιρίας. Αν δεν περάσει αυτή η συνθήκη θα καταρρεύσει όλη η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, το υπογράμμισε και ο εισηγητή. Η συνθήκη δεν είναι ιδανική, γιατί να την υπογράψουμε αν δεν είναι ιδανική. Μη βασίζεστε σε εμά για να το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, συγκεντρώσατε εδώ την αφρόκρεμα για να μιλήσετε για την υπογραφή αυτής της συνθήκης. Τίποτα δεν καταφέρετε καταφέρατε. Είμαστε στον ίδιο σχηματισμό, στο ίδιο υπόβαθρο με την TTIP. Επί της ουσίας δεν θα υπάρχει συμφωνία με τους λαούς. Εδώ καλέσατε εμπειρογνώμονες που είναι μόνο υπέρ της συνθήκης, υπέρ της συμφωνίας. Και στη συνέχεια αυτή η συμφωνία, αυτή η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ πριν προλάβουν να την ψηφίσουν τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν υπάρχει τίποτα το δημοκρατικό, αλλά και τίποτα το καινούριο στην πρακτική σας. Και αυτό βεβαίως θα ενθουσιάσει, θα συμπαρασύρει τα πλήθη άλλη μια φορά που περιμένουν από εμάς, νομίζετε εσείς, να ψηφίζουμε νόμους, ενώ στην ουσία περιμένουν οικονομική ανάπτυξη. Λόγω του κόστους παραγωγής που είναι μεγαλύτερο κατά 40% των Γάλλων εκτινοτρόφων βόλου και χοιρινού κρέατος θα υπάρξει μεγάλο πλήγμα ε, στη γαλλική οικονομία. 50.000 θέσει απασχόληση θα χαθούν στη Γαλλία, 200.000 θέσει απασχόληση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που το κόστο παραγωγή βόλου και χοιρινού κρέα είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ευρώπη από ότι είναι στον Καναδά. Ουσιαστικά εκχωρούμε την κληρονομιά μα στο βωμό των ελεύθερων συναλλαγών. Έχω μια τελείω διαφορετική αντίληψη από εσά για τη συνθήκη, για τη συμφωνία αυτή και έχω ένα ερώτημα να απευθύνω στο Γενικό Γραμματέα τη ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ. Για το μέλλον της γεωργίας, δεν πιστεύετε ότι θα είναι αρνητικός ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη και στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύετε ότι θα υπάρχει ε, απώλεια θέσεων απασχόλησης και μείωση των κερδών. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία χρειάζεται πράγματι αυτή τη συμφωνία σήμερα, τη συνθήκη σήμερα, ενώ διατρέχει μια περίοδο έντονης κρίσης. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχω και τέσσερα άλλα αιτήματα ε, παρεμβάσεων. Πέντε, έξι, εφτά. Και θα κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Αγαπητοί συνάδελφοι, τότε πρέπει να δώσω ένα λεπτό στον καθένα σας αφού είστε τόσο πολλοί. Η Καρολίν, ο Εμμανουέλ, η Αλέσια, ο κύριος Μάιερ. Μισό λεπτό να φτιάξω τον κατάλογο των ομιλητών. Οκτώ συνολικά, ένα λεπτό ο καθένας. Η Μαρία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εν συντομία, ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο της Κόπα Κοζέκα. Πώς εκτιμάτε την άποψη των μικρών αγροτών και γεωργών, Γάλλων, Γερμανών, ε, Ρουμάνων. Έχω δώσει σχετικά άρθρα στον τύπο που λένε ότι δεν τους εκπροσωπεί αυτή η συμφωνία. Ποια απάντηση δίνει η Κόπα Κοζέκα στο μικρό παραγωγό. Δεύτερο ερώτημα ε, στους αρχιτέκτονες. 500.000 αρχιτέκτονες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ελάχιστες είναι οι αρχιτεκτονικές επιχειρήσεις, ε, τα αρχιτεκτονικά γραφεία που ε, απαρτίζονται από περισσότερο από έναν ή δύο αρχιτέκτονες. Πόσους αρχιτέκτονες ε, αυτή τη στιγμή τους αφορά αυτό, το, αυτή, την εξαγωγη, αυτή η εξαγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή υπογράφουμε συμφωνία για 10 μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία ευρωπαϊκά που θα μπορούν να εξάγουν τις υπηρεσίες τους στο βωμό των υπολείπων. Και Τελικά στις 1600 σελίδες της ΣΕΤΑ δεν βρίσκεται κάτι τελείως διαφορετικό από την ερμηνευτική δήλωση 7 σελίδων ή είναι ε, νομικός δεσμευτική. Οι ασυνέπειες μεταξύ ε, κανονικής συμφωνίας και ερμηνευτικής δήλωσης πώς θα ρυθμιστούν και ποιος θα τις ερμηνεύσει όταν υπάρχουν αντιθέσεις στη διατύπωση. Όταν έχουμε επενδύσεις που... Ε, ε, που όταν έχουμε διατυπώσεις που είναι διαφορετικές, ποιος θα ερμηνεύσει το ένα κείμενο και το άλλο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι πρέπει κανείς να κάνει δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν είναι ιδανική η συμφωνία, αλλά είναι μια καλή συμφωνία. Είναι καλή, γιατί είναι τη δυνατότητα σε μια ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική να έχει προοπτική ώστε να διαμεσολαβήσει μεταξύ των συμφερόντων των μικρών και των μεγάλων. Ένα τεράστιο ποσοστό δασμών, ένα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, προστατευμένων ε, ονομασιών προέλευσης και μεταξύ μικρών και μεγάλων πρέπει να διακρίσουμε. Οι μικροί έχουν περιοχές προστατευμένες εσωτερικά. Οι μεγάλοι αναζητούν το διεθνές εμπόριο. Εγώ νομίζω ότι αν μια εμπορική πολιτική μπορεί να υφίσταται και πρέπει να υφίσταται, δεν μπορεί χωρίς μια τέτοια συμφωνία. Και επομένω σε πολιτικό επίπεδο ή πρέπει να υποστηριχθεί απολύτως αυτή η συμφωνία και ως προς το ρόλο της ε, Επιτροπής ή από ό,τι κατανοώ δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη συμφωνία που θα μπορούσε να υποστηρίξει κανεί. Και επομένω δεν θα είχαμε καμία συμφωνία και δεν θα είχαμε κανένα ρόλο να διαδραματίσουμε. Η Νεροντρίγιας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου αυτού οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο και έχουν κάνει παρουσίαση των απόψεών του. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα προ την Κομισιόν γιατί κάποιοι στρατηγικοί τομείς σε ό,τι αφορά την προστασία της αηφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος όπως είναι η εξόριξη ορυκτών, μεταφορές και ενέργεια δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία. Επίσης θα ήθελα να ξέρω γιατί ενώ είναι θετικό να υπάρξει η αμοιβαία αναγνώριση ε, σε εκπαιδευτικό επίπεδο υπάρχουν πολλές γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί. Μόνο 27 121 που αναγνωρίζουμε στη χώρα μου είναι μέσα στη συμφωνία. Σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση και επίσης υπάρχει μια πρόοδος σε ό,τι αφορά το άνοιγμα για τις δημόσιες προμήθειες με το να υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν υποεθνικές οντότητες αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αναγνώριση όλων των τίτλων που έχουν να κάνουν με, την, με τον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό θα είναι χρήσιμο περισσότερο σε επιχειρήσεις από τις επαγγελματίες του τομέα αυτό. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ το πρώτο σχόλιο μου. Είναι προς τους συναδέλφους. Πιστεύω την έλλειψη σεβασμού να απορρίπτεται τις ανησυχίες νομικών εμπειρογνωμόνων και μελών του Κοινοβουλίου ως φαντασιώσεις, ως φαντασιακές ανησυχίες. Δεν βοηθάει αυτό να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για την ε, ΣΥΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου συνδέεται με την ερμηνευτική δήλωση. Εάν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για τους διεθνείς επενδυτές, όπως είπε ο Ντέιβιτ, σημαίνει αυτό ότι περιορίζουμε το κεφάλαιο των επενδύσεων μόνο στις εθνικές επενδύσεις και έρουμε την και ε, αντιμετώπιση των επενδύσεων ανεξάρτητα από κάτω μέλος. Η Business Europe μας είπε ότι δεν θέλουμε περισσότερα δικαιώματα. Μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε να είσαστε ισότιμοι με τους εθνικούς επενδυτές και μήπως αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας και όχι μόνο σε μια ερμηνευτική δήλωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις μία για τον κύριο Πέσονεν. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα από τον Καναδά που, θα, που είναι απαγορευμένα στην Ευρώπη, ενώ ο Καναδά χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο γενετικά τροποποιημένους οργανισμού. Θεωρείται ρεαλιστικό ότι παρά την ΣΥΤΑ δεν θα έρθουν καθόλου γενετικά προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στο, στο πιάτο μα και στην κυρία Ρένσο. Μιλάτε για εναρμόνιση των προτύπων μέσα από τη ΣΥΤΑ και παρόμοια ε, προστασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Αλλά αυτό δεν βλέπω να γίνεται στο τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Εμείς έχουμε την αρχή της πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προτείνεται περισσότερο η Αμερικανική οδός, η οποία είναι πιο ταχεία και πιο απλή για την έγκριση των προϊόντων. Δεν θα οδηγήσει αυτό σε μια σύγκρουση οι δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις που θα πρέπει να επιληθεί σε νομικό, ερώτημα, σε νομικό επίπεδο. Και το τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο εισηγητή. Λέτε ότι οι συμφωνίες ευνοούν τους φτωχότερους. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Ναι, σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση για την κυρία Μελένα. Ποια είναι η επιστημονική βάση και η ενδείξη των μελετών επί των οποίων σήμερα μας εξέφρασε αυτή την ανησυχία σχετικά με την αύξηση των τιμών των φαρμάκων, των φαρμακευτικών προϊόντων. Και πώς μπορεί να καταδειχθεί ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο επί των ευρωπαϊκών τιμών αντίστοιχα. Δηλαδή, επί ποια βάση μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θα έχουμε αύξηση παθολογικών φαινομένων μέσω δηλαδή αυτής της συμφωνίας όπως είπατε. Ähm, Σας ευχαριστώ. Είναι μια σημαντική συμφωνία αυτή. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Από πολλές μελέτες ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό είναι απόλυτα θεμητό να διαφυσβητήσει κανεί ορισμένα σημεία. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Είναι κάποιε ανησυχίε όμω οι οποίε πρέπει να ληφθούν στα σοβαρά. Πιστεύουμε Ε, και το ψήφισμα για την TTIP που περιλαμβάνει μερικά σημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα και για την ΣΥΤΑ επίσης αυτή η ερμηνευτική δήλωση πώς μπορεί να συνάδει με αρχές όπως είναι η αρχή της ε, πρόληψης και πώς αυτό θα προστατεύσει τα πρότυπά μας και επίσης ποιοι είναι οι μηχανισμοί κυρώσεων λένε ορισμένοι ότι όλα αυτά βρίσκονται στη συμφωνία, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ασφα... ασαφής ο μηχανισμός για τις ε, κυρώσεις και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν τα πρότυπα. Μήπως θα ήταν καλύτερο λοιπόν όλα αυτά να βρίσκονται στο κείμενο της συμφωνίας και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων που να περιλαμβάνει και αυτά τα βασικά στοιχεία τα οποία τόνισαμε εμεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέλ. Νομίζω ότι η Σκά μίλησε για κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Ο συνάδελφος Ζωζέ Μποβέ έχει μπλοκαριστεί στον Καναδά και απειλείται με απέλαση γιατί πήγε να υπερασπιστεί τις ιδέες του για τη συνθήκη αυτή. Θα ήθελα να μας καθησυχάσετε γιατί είναι κάτι που θα πρέπει να προεβληματίζει όλους μας. Σε κάθε περίπτωση η συνθήκη αυτή είναι αμφίσιμη Πάρα πολλοί μας λένε ότι το, ο, ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι εξαιρετικά θετικός ή κάπως θετικός, γιατί άλλες οικονομικές μελέτες λένε ότι δεν θα είναι και τόσο σπουδαίος. Σε κάθε περίπτωση έχω μια ερώτηση για τον εκπρόσωπο της Κόπα Κοζέκα σε σχέση με το Brexit. Οι ποσοστώσεις βοήου και χοιρινό κρέατος έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει πώς αυτό θα πλήξει ή θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Γεωργία που, και ατροφία βέβαια που χυμάζεται κιόλα. Σε κάθε περίπτωση Υπάρχει ερμηνευτική δήλωση για ε, τη δημόσια υπηρεσία, το δημόσιο τομέα. Είναι ένα επιχείρημα που θα κάμψει ε, τις ανησυχίες των συναδέλφων που, ε, και τα λοιπά. Όμως παραμένει το ερώτημα. Όταν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του κειμένου της συνθήκης και του κειμένου της ερμηνευτικής δήλωσης, ποιο κείμενο θα υπερισχύσει. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους εμπειροχνόμονες. δύο λεπτά ο καθένας. Στη συνέχεια το λόγο θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν ο πρέσβης Κοστέλο του Καναδά και τέλος ο εισηγητής. Κύριε Πέσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σε ό,τι αφορά στη γεωργική κοινότητα και την πρόσβαση στην αγορά, είπα ξεκάθαρο ότι εν δυνάμει υπάρχει κίνδυνος διατάραξη αγοράς στον κλάδο του βόλου και χοιρινού κρέατος. Ας μην αποφύγουμε αυτή την παραδοχή. Ωστόσο, ω μέρος συνολικής συμφωνίας μπορούμε να το δεχθούμε εάν αυτοί οι δύο κλάδοι γίνουν αντικείμενο πραγματικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και μας ενδιαφέρει να γίνει σωστή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστό στο Καναδά στην αγορά γαλακτοκομικών. Είναι διαφορά, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Δεν εξάγουμε τα προβλήματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χτίσει τύχη ε, στην γαλακτοκομική αγορά. Γνωρίζουμε την οδυνηρή πραγματικότητα, ειδικά μετά το ρωσικό εμπάργο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ δραστήριος ε, εμπλεκόμενος φορέας στις συζητήσεις Ρωσίας-Ουκρανίας για την Κρυμαία. Οι Ευρωπαίοι Γεωργοί πλήρωσαν το τίμημα και ελπίζουμε ότι εσείς θα δουλέψετε έτσι ώστε να έχουν εναλλακτικέ αγορές οι Ευρωπαίοι Γεωργοί και κτηνοτρόφοι να ανοιχτεί η πρόσβαση προς την καναδική αγορά. Βεβαίως οι όγκοι της καναδικής αγοράς δεν αποκαθιστούν τις απώλειες που είχαμε από την απώλεια της ρωσικής αγοράς και αυτό το λέω εθνικά μιλώντας, παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτώ συλλογικά και να πω ότι στηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα ανοίξει μια εναλλακτική αγορά για τα υψηλής ποιότητα προϊόντα της Ευρώπης. Να πω ότι η διαχείριση και των εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των εξαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων λαμβάνει υπόψη ε, την ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν στη διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων και βεβαίως στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εγχείρημά της και πιέζουμε να ολοκληρωθεί ε, και πιέσαμε πολύ στο τελευταίο ε, κύκλο των διαπραγματεύσεων για να ενσωματωθούν όλα αυτά στο κείμενο. Ως προς τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς δεν υπάρχει καμία παρέκκληση από την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή καναδική νομοθεσία. Δεν πιστεύουμε ότι θα ε, επηρεαστεί το εμπόριο ε, γενετικό τροποποιημένων οργανισμών ε, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή και ό,τι να κάνει με τις ποσοστώσεις εισαγωγών, εξαγωγών και το Brexit φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα κατά πόσο θα υπάρχει συνολική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικεφαλής, έχει αναλάβει το καθήκον του καθορισμού των δασμολογικών ποσοστώσεων Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε συγκεκριμένες λύσεις ε, για συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, γιατί έτσι θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για να έχουμε πολλά και, πολλές και διαφορετικές ρυθμίσεις ανά περίπτωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια συνολικά για το θέμα. Η κυρία Σάντος, σας ευχαριστώ. Ήδη έχω παρουσιάσει κάποια παραδείγματα ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν πρόσβαση στην καναδική αγορά. Όταν ε, ε, πληρώνει κανείς 18% δεσμό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι ανταγωνιστικό στην καναδική αγορά ή σε όποια άλλη αγορά. Δεν είναι τεράστια αγορά θα μου πείτε. Ναι, αλλά αν δείτε όλες τις άλλες συμφωνίες και είναι πολλές, οι περισσότερες δεν πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας, να υπάρχει θετικό προηγούμενο και αν αυτή η συμφωνία δεν λύσει όλα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά, έστω. Θα λύσει όμως, θα βελτιώσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάποιες αγορές. Τώρα, για τις επενδύσεις και την προστασία των επενδυτών. Γνωρίζετε πολύ καλά τη θέση μας. Ως Business Europe δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το τωρινό σύστημα επίλυσης και διακανονισμού ε, διαφορών Η δυνατότητα των επενδυτών να προσφύγουν σε αυτό το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε μηχανισμό διακανονισμού διαφορών, γιατί υπάρχουν υποχρεώσει που απορρέουν από τη συνθήκη. Ε, πολλές είναι οι αμφιβολίες μας κατά πόσο τα εθνικά δικαστήρια θα ε, εφαρμόσουν ε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Για παράδειγμα, υποχρεώσεις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία θα είναι τα εθνικά δικαστήρια αρμόδια ε, που αφορούν καναδικές εταιρείες. Ε, Επομένω, καλύτερο είναι το σύστημα που προτείνεται. Ευχαριστώ. κύριος Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τον αριθμό των αρχιεκτών που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από τη δυνατότητα εξαγωγή των υπηρεσιών τους. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει με ακριβή επιστημονικό τρόπο. Ε, πάντως εξετάσαμε τη σταθερή ροή μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ με τη βάση τη συμφωνίας του 2008 που κάλυπτε τις ε, υπηρεσίες των επαγγελματιών. 175 περίπου γραφεία έχουν εγκατασταθεί στο Κεμπέκ αλλά γενικώ μιλώντας για την επαγγελματική κινητικότητα, ενώ εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί πολύ η κινητικότητα αυτή γιατί δεν υπάρχει δουλειά στην ουσία, έχει αυξηθεί προς τα έξω, εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι μελέτες λένε ότι περί το 8% των επαγγελματιών είναι κινούνται, μετακινούνται. Μάλιστα. Η κυρία Κλάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι η ΣΥΤΑ δεν θα τα επιτύχει όλα. Ξέρουμε ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε το εμπόριο, σε τι θέλουμε να εμπορευόμαστε και σε τι όχι. Και όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, έχουμε δει εκθέσεις για παράνομο εμπόριο πολύτιμων λίθων, ε, για βασανισμούς, ε, ε, έχουμε αποκλήσει συγκεκριμένες στα πλαίσια της ΓΚΑΤ από τους κανόνες του ΠΟΕ, ISDS θέλουμε να δημιουργήσουμε παγκόσμιο κανόνα. Στην πραγματικότητα όχι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον παγκόσμιο κανόνα του να μην υπάρχει κανόνας. Επομένως όλα εξαρτώνται από το είδο του εμπορίου και το είδο του κανόνα. Και για την Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει κανείς να αξιολογήσει με ανοιχτό μυαλό τα υπέρ και τα κατά ε, τη συμφωνία αυτή. Η ισορροπία στο τέλο εμεί θεωρούμε ότι δεν είναι και τόσο καλή. Ο ισολογισμό. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, κρίση στην υγεία και την λιτότητα στην υγεία. Και νομίζω ότι και εδώ μπορεί να βοηθήσει η συζήτηση αυτή, γιατί χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις, ώστε να έχουμε βιώσιμε υπηρεσίες και στο πεδίο αυτό. Και αν, δεν, αν μου επιτρέπει ο γείτονά μου, ε, το 40% της δουλειάς των αρχιεκτόνων είναι στις δημόσιες ε, συμφωνίες, συμβάσεις. Επομένως, σε ό,τι αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. Θα έλεγα λοιπόν το εξή. Υπάρχουν προβλήματα στη ΣΥΤΑ. Αν δεν θεωρείτε ότι ε, ενέχει προβλήματα η συμφωνία, τότε η δήλωση δεν έχει κανένα νόημα. Αν θεωρείτε ότι ναι, έχει κάποια προβλήματα, πρέπει να δούμε κατά πόσον η δήλωση αυτή μας βοηθάει να τα καλύψουμε. Αυτό είναι ε, το καθήκον που έχουμε μπροστά μα. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί πώ μια δήλωση μπορεί να αντικαταστήσει τμήματα του κειμένου που δεν συνετάξαν ποτέ. Αυτά που λέει πρέπει να εξισορροπούνται με αυτά που δεν λέει. Κανείς δεν είπε ότι η ΣΥΤΑ ιδιωτικοποιεί τις κυβερνήσεις. Το να το βάλουμε σε μια δήλωση δεν θα βοηθούσε. Αυτό που θα βοηθούσε είναι ότι η ΣΥΤΑ δεν υποσκάπτει την νομοθεσία τις νομοθετικές διατάξεις. Ευχαριστώ κύριε Αρένσο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ υποστηρίζω τι εκκλήσει πολλών μελών της Επιτροπής σα να διαμφισβητήσουμε τη νομική βάση αυτής τη ερμηνευτικής δήλωση. Δεν ξέρουμε πόσο νομικά δεσμευτική είναι, αν θα τη λάβουν υπόψη οι δικαστέ αν υπάρξει κάποια νομική προσφυγή. Χαιρετήσουμε την δήλωση ότι αναγνωρίζονται και οι ανησυχίες της κοινή γνώμης και αυτό είναι κάτι χωρίς προηγούμενο ότι θα πρέπει να εμπλακεί και η κοινή γνώμη. Σίγουρα αυτό δεν ίσχυσε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του κειμένου αυτού καθεαυτού. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική η δήλωση. Απλώς δείχνει ότι οι διαπραγματευτές καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί πολλές ανησυχίες στο κείμενο της συμφωνίας για την προστασία των επενδυτών λέει ότι επιτρέπεται να υπάρχουν συστήματα για, την, για, για διαιτητικές λύσεις για να αποφευθούν παραπλανητικές αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε, το να τροποποιηθεί αυτό αργότερα και να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε δυσκολία στα, στη συμφωνία αργότερα. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ πραγματιστικό ούτε αξιόπιστο. Πώ θα λειτουργήσει λοιπόν αυτό στο μέλλον. Και τονίζω και πάλι ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα νομικά προβλήματα για την διαιτησία σε διαμάχες επενδύσεων και κρατών που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Ένωση των Γερμανών ε, Νομομαθών ζήτησε να υπάρξει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ κέριο να το κάνουμε αυτό τώρα και να διευκρινιστεί και να μην έχουμε πολλά χρόνια νομικών διαμαχών, ιδίω για τι ρήτρε προστασία επενδυτών. Και για το αν είναι πιο προσφυσιτέ ή λιγότερο οι υγειονομικέ υπηρεσίε και αν θα έχουμε περισσότερα βλαβερά προϊόντα και περισσότερες ασθένειες και για την τιμή των ε, φαρμάκων θα ζητήσουμε να υπάρχει μια έκθεση αντικτύπου και από τις δύο πλευρές ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες ε, προετοιμασίες αν χρειαστεί να καλύψουν κάποιες ζημίες που θα προκύψουν από τη συμφωνία. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, γιατί αλλιώ ούτε μέχρι το βράδυ δεν προφθαίνω. Κάποια βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, οι ανησυχίε που ακούσαμε σήμερα και έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, τις παίρνουμε πάντα στα σοβαρά αυτέ τι ανησυχίε Γι' αυτό τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε αυτή την ε, ε, άσκηση του να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το να λάβουμε υπόψη αυτέ τι ανησυχίε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατρέψουμε τη θεσμική διαδικασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν διαπραγματεύεται μία συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα και ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, τις έχουμε λάβει υπόψη αυτές τις ανησυχίες. Τώρα εναπόκειται στο Συμβούλιο να συνάψει τη συμφωνία με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε αν είναι καλή ή όχι αυτή η συμφωνία, είναι επαρκής. Εμείς την έχουμε διαπραγματευτεί, τέρμα η διαπραγματεύση. Και τώρα θα πρέπει να δούμε αν αυτή η συμφωνία είναι καλή ή όχι για την Ευρώπη και για τον Καναδά λοιπόν Φυσικά, αλλά αυτό, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Το λέω αυτό γιατί η κοινή δήλωση είναι μια ερμηνευτικού χαρακτήρα δήλωση. Δεν αλλάζει τη μορφή τη συμφωνία, δεν έχει στόχο να αλλάξει η συμφωνία. Και είμαστε πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της δηλώσεως και του περιεχόμενου της συμφωνίας. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε απλή γλώσσα, σε απλά αγγλικά και ενδεχομένω σε όλες τις ευρωπαϊκές επίσημες γλώσσες αυτά που εκφράζονται νομικά στην συμφωνία. Για να σταθώ μονάχα σε μία από τις ανησυχίες της δημόσιας υπηρεσίας. Έχουμε ακούσει από την Ένωση των Δημοσίων Υπηρεσιών ότι η ΣΥΤΑ οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Όχι, δεν το κάνει. Μπορούμε να σας δείξουμε και τις τρεις σελίδες των νομικών αναφορών που δείχνουν γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω που είναι οι ρήτρε που δείχνουν ότι η ΣΥΤΑ οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση. Αν έχετε όμω αμφιβολίε, σα το λέμε αυτό και σε απλή γλώσσα στην ερμηνευτική δήλωση. Δεν εμποδίζει το να παραμείνει στο δημόσιο τομέα οι δημόσιε υπηρεσίε, αν όμω αν κάποιος Δήμος ακολουθεί την των ιδιωτικών υπηρεσιών και μετά δεν ικανοποιημένο. Μπορούμε να το δείξουμε και από την νομική ανάλυση. Δεν περιμένουμε ότι ο κάθε πολίτης θα είναι εμπειρογνώμων στο διεθνές δίκαιο. Το λέμε αυτό σε απλή γλώσσα. Η ΣΥΤΑ δεν εμποδίζει τις δημόσιες αρχές από το να επαναδημοσιοποιήσει, να, να κάνει δημόσιες πάλι υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Επίσης, η αξία αυτής της δήλωσης, εγώ μπορώ να σας δώσω μια επίσημη δήλωση γιατί βάσει της ε, Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συμβάσεων έχει νομική αξία αυτή η συμφωνία. Εμείς έχουμε καταφέρει να φέρουμε από κοινού τη νομική υπηρεσία της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Καναδά. Και αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα. Και οι υπηρεσίες του Συμβουλίου τόνισαν ότι είναι μια ερμηνευτική ε, δήλωση. Είναι, είναι νομικά δεσμευτική αυτή η δήλωση. Όπως το βλέπουμε εμείς, ένα δικαστήριο θα ερμηνεύσει εάν έχει αμφιβολίες για το κείμενο της ΣΥΤΑ, για την ερμηνεία του κειμένου, θα έπρεπε να ακολουθήσει την ερμηνευτική διάταξη. Δεν έχει τελειώσει η συζήτηση. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να προκύψει μια τελική μορφή του κειμένου, αν υπάρξει και η απόφαση του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα, αλλά εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες και επεξεργασία για θέματα τα οποία δεν είναι ίσονος σημασίας κάτι ακόμα για να διαλύσω να διώξω κάποιες παρεξήγησεις για τα θέματα αυτά. Δημόσιες υπηρεσίες, νερό, υγειονομική περίθαλψη, παιδεία. Συγγνώμη, εδώ πέρα σεβόμαστε τι δημοκρατικέ επιλογέ των κρατών μελών μα. Κάποια κρατημέλη μα έχουν ε, ιδιωτικοποιήσει αυτέ τι υπηρεσίε εν μέρη ή πλήρω. Αυτό είναι δική του υπόθεση, είναι δικαίωμά του. Εφόσον δεν αλλάζουν <clears throat> την άποψή του, έχουμε μια δημόσια μια κοινή αγορά όπου οι δημόσιες και ιδιωτικές ε, υπηρεσίες βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και επί τη βάση αυτού κάνουμε τις συμφωνίες. Αν όλα τα κρατημέρια ξαναφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο τομέα, η ΣΥΤΑ δεν θα τους εμποδίσει και οι ξένοι επενδυτές δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Το δικαίωμα ρυθμίσεις. Και πάλι είναι πάρα πολύ σαφής η ερμηνευτική δήλωση. Και η συμφωνία είναι πάρα πολύ σαφής δεν παραχωρούμε το δικαίωμα ρύθμισης στην Ευρώπη. Το δικαίωμα τη ρύθμιση στην Ευρώπη δεν είναι η άδεια να κάνει κανεί οτιδήποτε. Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί για το δικαίωμα ρύθμισης που υπάρχουν και στα συντάγματά μας. Δεν έχουν το δικαίωμα οι ρυθμιστές να αποφασίσουν για τα πάντα στην ανθρώπινη ζωή. Ακολουθούν κάποιου κανόνε και οι κανόνες τη ΣΥΤΑ σέβονται απόλυτα τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δικαίωμα της ρύθμισης και σε καθένα από τα κρατημένη μας. Κάτι ακόμα. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Όχι, δεν θα υπάρξουν προϊόντα γενετικά τροποποιημένα τα οποία δεν εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα εισαχθούν προϊόντα από τον Καναδά που δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Η αρχή της πρόληψης είναι μια σημαντική αρχή, περιλαμβάνεται στην ε, συνθήκη αυτή η Κομισιόν δεν θα παραβιάσει την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδάς το κατανοεί αυτό. Ακόμα και πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων υπήρξε μια πολιτική συμφωνία με τον Καναδά ότι δεν θα αναδιαπραγματευτούμε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Γιατί εκεί θα είχαμε πει όχι, δεν θα διαπραγματευτούμε και το ίδιο αφορά το κρέας το οποίο έχει περάσει επεξεργασία με ορμόνες κτλ. Γεωγραφικές ενδείξεις δεν έχουν διεθνές εμπόριο με τον Καναδά όλα τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτά τα οποία έχουμε είναι μια επιλογή αυτών που έχει γίνει από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν δεν έχει απορρίψει ούτε μία αίτηση κράτου μέλου για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη. Πολλές φορές έχουμε έχουμε δει αιτήσει για να τροποποιείται ο, ο κατάλογος και έχουμε και μερικά στοιχεία γεωγραφικής προέλευσης που μπήκαν τελευταία στιγμή. Αν λοιπόν το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη ό,τι θέλουν το έχουμε στη συνθήκη. Δεν ξέρω από πού προέρχονται οι προτιμήσεις των κρατών μελών, αλλά ρωτάνε, και αυτό είναι λογικό, αν υπάρχει εμπόριο σε αυτά τα προϊόντα. και αυτό αντανακλά λοιπόν ο κατάλογος γεωγραφικών προελεύσεων είναι μια σωστή κατά την άποψή μου απεικόνηση του τι εμπορευόμαστε με τον Καναδά. Μπορεί κάποιο στο μέλλον να θέλει και ένα πρόσθετο προϊόν το οποίο πρέπει να απελευθεί στον κατάλογο, αλλά μέχρι όπου μέχρι την ε, σύναψη της ε, συμφωνίας ΣΥΤΑ, ο Καναδάς ήταν εναντίον της ιδέας της γεωγραφικής προέλευσης. Έχουμε πείσει λοιπόν τον Καναδά να ακολουθήσει ένα σύστημα sui generis το οποίο αντανακλά και το ευρωπαϊκό σύστημα. Αρχίσουν και οι επαρχίε του Καναδά να έχουν τα δικά του συστήματα γεωγραφικής προέλευσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας λογικής συζήτησης με τον Καναδά. Δεν λέω ότι ο Καναδάς θα μας ακολουθήσει απόλυτα στον τομέα αυτό, αλλά δεν ήταν εύκολο να τους πείσουμε να δεχτούν ένα σύστημα που μοιάζει με το δικό μας. Κάτι ακόμα για την αξία αυτής της συμφωνίας άμα δείτε τα μακροοικονομικά συστήματα, οτιδήποτε είναι μικρό σε σχέση με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξαγωγής. Μιλάμε για δισεκατομμύρια σε εξαγωγές, χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες θα κερδιθούν. Δεν υπάρχει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποια μελέτη που λέει ότι θα υπάρξει απώλεια θέσεων απασχόληση και δεν υπάρχει ακόμα μια επίσημη άποψη Κομισιόν για τι συνέπειε στην απασχόληση συμφωνία. Το επεξεργαζόμαστε ακόμα. Για τον Ντέβιτ, ε, για την αηφόρο ανάπτυξη. Ναι, μα είναι δεσμευτική η αρχή αυτή. Δεν έχουμε κυρώσει. Αλλά αυτή είναι και η ομόφωνη <clears throat> θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη-μέλη είναι ομόφωνα για αυτό το θέμα και το Κοινοβούλιο επίσης γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν οι εμπορικές κυρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι των αναπτυσσομένων χωρών για παραβίαση εργασιακών αρχών. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση για το αν πρέπει να αλλάξει αυτή η προσέγγιση και θα είναι μια δύσκολη συζήτηση που δεν μπορούμε να την αλλάξουμε σε μια συζήτηση τη ρήτρα που υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα ξανανοίξουμε το θέμα αυτό με τον Καναδά και θα το επανεξετάσουμε και μέχρι τότε ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στην Ευρώπη αν θέλουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση μας ή όχι. Αν θέλουμε να έχουμε εμπορικές ε, κυρώσεις για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων. Αν είναι αυτό η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να υπάρχουν αυτά. Τέλος, είπε κάποιος ότι οι ευρωπαϊκές συμφωνίες δεν καλύπτουν τα πάντα. Φυσικά δεν μπορούν να θεραπεύσουν όλα τα κακά του κόσμου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και δημιουργούν πλούτο. Δεν μπορούν όμως να εγγύθουν μια ισοδίκαια κατανομή του πλούτου. Εμείς ως ε, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς ως κοινοβουλευτικοί, εσείς θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει ισοδίκαια διανομή των κερδών από αυτή τη συμφωνία το Διεθνές Γραφείο Εργασίας εξασφαλίζει την εξάλληψη των δασμών. Όχι. Ασχολείται με τα εργασιακά δικαιώματα. Εμείς ασχολούμαστε με το εμπόριο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό σύνδεσης με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και αυτό είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουμε. Δεν είναι κάτι που το έχει αρνηθεί να το αναγνωρίσει ο καναδά στις βασικές αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Υπάρχει όμως ένα πολιτικό πρόβλημα με κάποιες από τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και η συμφωνία αυτή τους έχει βοηθήσει να αλλάξουν τη γνώμη τους. Δεν πρόκειται για μια συμφωνία σε εμπορικό επίπεδο και δεν είναι ο στόχος της να είναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και για το νομικά δεσμευτικό της ε, κοινή ε, δήλωσης, ερμηνευτικής δήλωσης. Ήταν ε, πολύτιμα αυτά που μας είπατε βάσει του 31 της Σύμβασης της Βιέννης, λέτε, θα το ελέξει και η δική μας νομική υπηρεσία. Αλλά για, πιστεύω ότι αυτό είναι από τα κέρια θέματα πρέπει να μας απασχολήσει το αν είναι νομικά δεσμευτική ή όχι αυτή η ερμηνευτική δήλωση. Και η δήλωση αυτή είναι κομμάτι της συνολικής συμφωνίας. Καλά λέει ο πρόεδρος. Κύριε Πεσβευτά, έχετε παρακολουθήσει αυτή τη θαυμάσια συζήτηση στην Επιτροπή μας και θα θέλαμε να έχουμε τη δική σας άποψη για τη συμφωνία αυτή. Είναι δύσκολο να μιμηθεί κανείς ε, τον ΟΟ ε, και είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε μια τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς δεν έχω απαντήσει για τα πάντα, αλλά επιτρέψτε μου κάποια σύντομα σχόλια. Ε, πιο ειδικά και πιο γενικά. Ελπίζω να καταφέρω να τοποθετηθώ μεταξύ του μεταφυσικού επίπεδου. Δεν θέλω να μιλήσω για το ρόλο του παραδείσου σήμερα. Και έχετε και την, με τον ε, Μάρο ε, έναν πραγματικό βιρτουόζο σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Λοιπόν, εμείς ε, σημειώνουμε και κατανοούμε τις ανασυχίες ε, των ε, Ευρωπαίων καλλιεργητών, των γεωργών, τις έχουμε και στον Καναδά. Ήταν μια δύσκολη περιοχή αυτή. Αλλά πετύχαμε. Πετύχαμε κάποια πράγματα. Κατανοώ αυτά που λέτε για τους κινδύνους. Αλλά η πρόσβαση της πιστώσης είναι κάτω από 1% της αγοράς του βοήου και λιγότερο από μισό του χοιρινού. Αντίστροφα για τους Ευρωπαίους καλλιεργητές η πρόσβαση είναι πολύ σημαντική στην καναδική αγορά. Επομένως αυτό ήταν για μας μια πολύ πολύ δύσκολη παραχώρηση. Ε, γιατί ε, ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους δικούς μας γεωργούς, που πολύ συχνά είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως και έχουν μεταφέρει τις δικές σας παραδόσεις, γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτές τις παραχωρήσεις. Τώρα για την κυρία Κρέντσο ε, κατανοούμε τις ανησυχίες σας, αλλά έχουμε την ίδια φιλοδοξία με εσά να προστατεύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες του Καναδά. Και είμαστε υπερήφανοι για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουμε στον Καναδά και θέλαμε να είμαστε απολύτως σαφείς. Θέλουμε να νομοθετήσουμε προς όφελος και προς το συμφέρον των δημοσίων υπηρεσιών και του επίπεδου που παρέχουμε στους πολίτες. Αλλά και πάλι επιβεβαιώθηκε σήμερα η, η πάγια θέση μου ότι δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ε, ως προς αυτό. Έχουν κυκλοφορήσει τώρα διάφορες ε, εκδοχές του κειμένου, ε, πρώιμες, ύστερες κτλ. Και ο τύπος έχει σχολιάσει. Όταν έχουμε την τελική, νομίζω ότι θα... Τελικώς θα έχει επιτύχει να υπερασπίσει και τις, τα συμφέροντα και των δύο, και των δύο πλευρών. Αυτό είναι προσπαθήσαμε να επιτύχουμε από την αρχή. και μέσω της συζήτησης του Υπουργού και του Πρωθυπουργού και από τις ενώσεις και τους φορείς που ε, επισκέφθηκαν τον Καναδά ε, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και ήταν καλοδεχούμενες αυτές τις συζητήσεις ε, για τις συλλογικές συμβάσεις, τις διατάξεις του ILO κτλ. Έχουμε δεσμευτεί για την επικύρωση αυτή. Αυτό όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα δυσκολίας αρμοδιότητας με τις ομοσπονδιακές ενότητες του Καναδά Αυτό έχει εγγραφεί στο ε, εργασιακό δίκαιο στον Καναδά αλλά χαιρετίζω τις παρατηρήσεις σας και για το πόσο επικοδομητικές υπήρξαν οι συζητήσεις αυτές. Έχουμε μάθει πολλά και εμείς και εσείς από αυτές τις συζητήσεις για τις θεωρήσεις ε, θα ξέρετε ότι τον περασμένο Ιούλιο είχαμε παράσχει ένα χρονοδιάγραμμα για την άρση των προϋποθέσεων και στην ουσία για την ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών στον Καναδά. Αυτό θα έχει επικυρωθεί πάρα πολύ σύντομα, αυτό μπορώ να πω σήμερα, και για μια συγκεκριμένη υπόθεση που αναφέρθηκε στον τύπο ε, δεν μπορώ να για λόγους ιδιωτικότητας ε, να σχολιάσω συγκεκριμένη περίπτωση αλλά οι συνάδελφοι το γνωρίζουν και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα για το θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να πω εδώ επίσημα ότι οι καναδικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, υποστηρίζουν ένθερμα την ΣΥΤΑ όπως είχαν κάνει και για την ΝΑΦΤΑ. γιατί έχουν δει τις ωφέλειες Ε, γιατί εμείς είμαστε μικροί εξορισμού. Δείτε τα μεγέθη εδώ πέρα που συζητούμε Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς. Ε, Όμω, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τον Καναδά υποστηρίζουν, ξαναλέω, ζεστά τη συμφωνία αυτή, όπω έκαναν και με άλλε. Γενικότερα, ήθελα να κάνω την εξή έκκληση. Πώ το βλέπουμε εμεί, οι Καναδοί, εμείς είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία, είμαστε πάντα υπέρ του εμπορίου. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο για τις ε, θέσεις απασχόλησης. Ε, χρειάζεται να έχουμε μια διαφοροποιημένη οικονομική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργό ε, Τρούντο εξελέγει για να προστατεύσει τη μεσαία τάξη. Μιλούμε για μια 20% αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μας με τεράστια κέρδη και για τι δύο πλευρές αυτά θέλουμε να μεταφραστούν σε ευημερία και περισσότερη προστασία για τη μεσαία τάξη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προοδευτική η συμφωνία αυτή. Ε, έχουμε δεσμευτεί για ένα ισχυρό ρόλο για την κυβέρνηση, για το κράτος, όπως και εσείς. Έχουμε κοινά κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα. Κάποιες φορές έχουμε διαφοροποιημένες επιλογές ενδεχομένως, αλλά θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο προοδευτική συμφωνία που υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο και οι εκπρόσωποι της κυβέρνηση είναι δεσμευμένοι προς την προώθηση αυτής της ατζέντα, αυτού του θεματολογίου διεθνώς, παγκόσμια. Αυτού του προτύπου των συμφωνιών. Και εμείς σκεπτόμαστε του πού πάει η παγκοσμιοποίηση και ποιες είναι οι ωφέλειες του εμπορίου, ότι πρέπει να είναι συμμετοχική η ανάπτυξη οικονομική που επιτυχάνουμε. Αυτά είναι για μας βασικές αρχές. Και, αυτή, και έτσι πλαισιώνω και την τη στρατηγική εξέταση του πού πάει ο κόσμος. Ναι, όμως ο κόσμος αλλάζει. Αναδύονται νέε δυνάμεις, οι ρόλοι αλλάζουν, ε, είναι δυναμικοί. Οι σχέσεις είναι δυναμικές. Και ε, συνεισφέρουμε όλοι στο να εγγράψουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, του διεθνούς παιχνιδιού, του εμπορίου. Και ξέρουμε ότι είμαστε σύμμαχοι και φίλοι σε αυτή την προσπάθεια εμείς και εσείς και μιλούμε για μια ευρύτατη σχέση σε πάρα πολλά επίπεδα και πολύ βαθιά. Ε, και αυτό που συζητούμε εδώ σήμερα δεν είναι τυχαίο, δεν προέκυψε έτσι ως ατύχημα. Γιατί βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα μπροστά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, ε, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την προστασία δικαιωμάτων των θεμελιωδών Νομίζω ότι και η ΣΕΤΑ και οι συμφωνίε και αυτή μας βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, οι διατάξεις για την κινητικότητα είναι πολύ σημαντικές. Και τέτοια πλαίσια συνεργασίας ε, ε, συνεισφέρουν στην ομαδοποίηση, στην κοινωνική συμμετοχικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι και λόγω της οικογένειας μου και της γυναίκας μου παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει όταν συνδυαζόμαστε οι με τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε πολλά από τα σχόλιά μας και αν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα βεβαίως μπορείτε να τα συζητήσετε διμερώς με τα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Στρέφομαι τώρα στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να κάνω δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Καταχάσα ε, τα ωφέλη για τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους φτωχούς. Εάν συνάψουμε αυτή την εμπορική συμφωνία και την εφαρμόσουμε αποτελεσματικά, η παραγωγή κλωστοϊφαντουργίας, για παράδειγμα στην Ινδονησία, θα μπορούν να πουλήσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Καναδά. Και ο Economist στην έκδοσή του από 3 μέχρι 7 Οκτωβρίου ε, έχει ένα άρθρο που εξηγεί ξεκάθαρα πώς οι φτωχοί ωφελούνται περισσότερο από μια διεθνή ε, συμφωνία, πολύ περισσότερο από τους πλούσιους. Σας παρακαλώ να το διαβάσετε γιατί έχει εκεί πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα συμφωνώ με τον κύριο Πέσονεν από τη Φιλανδία στα λεγόμενά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλώς υιοθέτησε τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας. Υιοθέτησε τις κυρώσεις όχι με οικονομικό γνώμονα, αλλά με γνώμονα τις αξίες της. Η Φιλανδία και άλλες χώρες περιμένουν λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να δώσει εναλλακτικέ, να ε, προσφέρει εναλλακτικέ αγορές. Και πού θα τις βρει ε, αν δεν είναι χώρες με ίδια νοοτροπία με εμά όπως είναι ο Καναδάς. Για κάποιους από εμάς η απόφαση για τη ΣΥΤΑ δεν είναι θέμα γεγονότων και ε, ε πραγματικοτήτων. Είναι θέμα ιδεολογικής διαμάχης. Ως προς την κοινή δήλωση δεν έχει σκοπό να βελτιώσει τη ΣΥΤΑ γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτή καθε αυτή. Είναι ε, για να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Αν θέλει κανείς το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ε, τότε θα πρέπει αυτή τη γνώση να την παρουσιάσουμε με γλώσσα απλή. Και έτσι ερμηνεύω εγώ αυτή την ερμηνευτική δήλωση. Πάρα πολλοί θαυμάσιοι άνθρωποι από την πολύ άκρα δεξιά και την πολύ άκρα αριστερά, αν μου επιτρέπεται ο όρος, με χαρά λένε ότι δεν θέλουν να στηρίξουν τη ΣΥΤΑ γιατί δεν είναι μια συμφωνία που να δημιουργεί έναν ιδανικό παράδεισο. Ταυτόχρονος ευχαρίστως κάνουν εμπόριο με τις χώρες όπως είναι η Ρωσία χωρίς να θέτουν επιπρόσθετα ερωτήματα. Και αυτό ε, ισχύει και αληθεύει εάν δει κανείς και τη διατύπωση της επιχειρηματολογίας τους. Εμείς λοιπόν που έχουμε την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι έχουμε και την πλειοψηφία της κοινή γνώμης, θα υπερασπιστούμε τις αξίες της ανάπτυξης και της δικαιοσύνης και έτσι θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη του συντομότερων δυνατών. Σας ευχαριστώ. So, thanks a lot to rapporteurs, thanks a lot to our experts. Uh, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους εμπειρογνώμονες, όλους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ τον Μόρο και τον ε, πρεσβευτή και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες συζητήσεις σε επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. So, then we switch to um, point 6 and 7. Πάμε στα σημεία 6 και 7. Έχουμε μια κοινή συζήτηση τώρα για την ε, παράταση, των, την επέκταση μάλλον των διατάξεων συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με το Ουσμπεκιστάν στο διμερέ επίπεδο κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Καταλαβαίνω ότι θα φύγετε, αλλά και αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με εργασιακά δικαιώματα, με καταναγκαστική παιδική εργασία. Παρακαλώ, τουλάχιστον φύγετε σιωπηλά. Κοινή συζήτηση λοιπόν με το, για την εταιρική σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Θυμόσαστε ότι είχαμε αναβάλει τη συζήτηση αυτή για πολύ χρονικό διάστημα γιατί υπήρχαν περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας παιδιών στο Ουσμπεκιστάν για την συντομιδή ε, και ζητήσαμε από το, από το Οργανισμό Εργασίας να ελέγξει την κατάσταση και να μας αναφέρει αν υπήρχε κάποια βελτίωση στα θέματα αυτά. Συζητήσαμε και τον προηγούμενο μήνα και είχαμε και μια δήλωση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για το θέμα αυτό και τώρα έχουμε μια περαιτέρω συζήτηση και με την συγγήτριά μας τη Μαρία Αρένα για το θέμα αυτό και θα της δώσω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι, ότι το ζήτημα αυτό δείχνει ότι ορισμένοι δεν λειτουργούν ιδεολογικά και μόνο. Το 2011 θυμόσαστε ότι το Κοινοβούλιο <clears throat> είχε πάρει από το Συμβούλιο μια αίτηση νομοδότηση για τη συμφωνία αυτή με, για τα κλωστοεφαντουργικά. Το Κοινοβούλιο μετά ψήφισε μια έκθεση που αφορά τα θέματα τη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και το θέμα τη κλωστοεφαντουργίας ήταν κέριο σε ό,τι αφορά την καταναγκαστική εργασία και την προστασία των παιδιών. Το 2013 το 2013 συνεργάζεται με το Διεθνή Οργανισμό Εργασία στο Ουσβεκιστάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο και γι' αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η συνεργασία αυτή οδήγησε σε κάποιες επίτρο ε, αποστολές παρακολούθησης για να εποπτευθεί η συγκομιδή βάμβακος. Οι εκθέσεις λένε ότι σε ό,τι αφορά τα παιδιά έχει σχεδόν σταματήσει η χρήση παιδιών, αλλά η καναγκαστική εργασία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Υπάρχουν ενέργειες συνειδητοποίησης και προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες εργασία και έχει δεσμευτεί στο, πρόγραμμα, στο Decent Work Program υπό την αιγίδα του διεθνού ε, Οργανισμού Εργασίας. Υπήρξαν λοιπόν πρόοδοι σε ό,τι αφορά το θέμα τη παιδική εργασία και τη καταναγκαστική εργασία και οι βελτιώσει οι οποίε έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια τη συγκομιδή ε, Φάμβακο <clears throat> είναι και αποτέλεσμα μια θετική συνεργασία στην κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν με τον Διεθνή Οργανισμό εργασία. Πιστεύω ότι μετά από την ε, έκθεση αυτή θα πρότεινα να υπάρξει η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, τροπολογίες να εγκρίνουμε για αυτή τη συμφωνία για τα κλωστοϊφαντουργικά. Αυτό, αυτή η έγκριση συνδέεται με ένα ψήφισμα που ζητά από τι αρχέ του Ουσμπεκιστάν να συνεχίσουν εργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασία για να σταματήσει οριστικά η καταγαναγκαστική εργασία και να υλοποιηθεί η αξιοπρεπή εργασία στην συλλογή Βάμακο. Ζητούμε επίση από την Κομισιόν και μέσα από την τοπική αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει την εφαρμογή των κανόνων για την καταναγκαστική εργασία και σε περίπτωση κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί το Κοινοβούλιο να ενεργοποιήσει την ανασταλτική ρήτρα που αναφέρεται στο άρθρο 92 τη συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα και συνεργασία, είναι απαραίτητο να το υπενθυμίσω και αυτό, μέσα, Όπω θα γίνει μέσα στο ψήφισμά μα. Επίση, θα ακούσω με προσοχή τι παρατηρήσει των συναδέλφων και ιδίω των σκιεδών εισηγητών και περιμένω τις τροπολογίες σας για τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Οκτωβρίου. 19 Οκτωβρίου θα συναντηθούμε με την ομάδα παρακολούθησης. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα εκδώσει την γνωμοδότηση της στις 20 Οκτωβρίου, 9 και 10 Νοεμβρίου στην Αρμόδια Επιτροπή η ψηφοφορία και μετά πάμε στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι παρόν κάποιος σκιώδης εισηγητής, εσείς όμως αντικαθιστάτε κάποιον, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κρίστα Λορόβο, η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα, έχει κάποιο θέμα με την υγεία της, ωστόσο μου ζήτησε να μιλήσω για την επέκταση των διατάξεων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσμπεκιστάν στο ε, διμερές εμπόριο κλωστοϊφαντοργικών προϊόντων. Ευχαριστεί λοιπόν η κυρία Μαρία Αρένα, τον εισηγητή, και για την πρότασή του να επεκταθεί το πρωτόκολλο αυτό. Σα ζητώ να συμφωνήσετε με την πρόταση αυτή και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να ε, συγκατατεθεί. Θέλουμε να επεκτείνουμε αυτές τις διατάξεις για να υπάρχει συνοχή με την προηγούμενη επιχειρηματολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Το 2011 αρνηθήκαμε ε, την επέκταση, γιατί θεωρούσαμε ότι έπρεπε να υπάρχουν σε βάθος αλλαγές στο Ουσμπεκιστάν. Σήμερα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία ε, τρία έως πέντε χρόνια το Ουσμπεκιστάν άλλαξε και βελτιώθηκε σημαντικά ε, στον τομέα της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας. Πράγματι μένει απόσταση να διανυθεί και αυτό το αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οφείλει να αναγνωρίζει και τις τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει το Ουσμπεκιστάν. Η βελτίωση των ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι βαθμιά σταδιακή, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια νύχτα. Με την έκριση αυτού του πρωτοκόλου στέλνουμε θετικό μήνυμα και καλούμε το Ουσπεκιστάν το παροτρύνουμε, να βελτιώσει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα κίνητρο για πρόοδο στη χώρα αυτή γενικότερα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες στη χώρα αυτή. Άρα Έχουμε έτσι μια ευκαιρία. Ε, καθιστάμεθα χρήσιμη. Έχουμε την ευκαιρία να βελτιωθεί κάτι έξω από τα σύνορά μας. Όταν βλέπει κανείς αυτό που συμβαίνει στο Ουσπεκιστάν διαπιστώνει ότι στις 22 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος ε, υπόγραψε έναν αναθεωρημένο νόμο για τις εργασιακές σχέσεις που τηρεί τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και τα δύο τμήματα ε, της Βουλής ενέκριναν αυτό το ε, νομοσχέδιο, ενώ το Κοινοβούλιο θα κυρώσει τη σχετική συνθήκη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σήμερα, σύμφωνα με την ε, συμφωνία μας. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δείχνουν ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο Ουσβεκιστάν και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό χάρη στις δικές μας διαπραγματεύσεις. Δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα ως προς την κατεύθυνση που έχουν ε, ε, έχουν επιλέξει οι πολιτικοί στη χώρα αυτή. Η κυρία Σάρκη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη ο Χάνου Τάκουλα δεν μπορούσε να είναι παρόν. Θα διαβάσω απλώς το κείμενο το οποίο έχει προετοιμάσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που η Επιτροπή μας είναι έτοιμη να προχωρήσει για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα έργο από το 2011 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ανανέωσε το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ουσμπεκιστάν. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Αρένα για το καλό της σχέδιο έκθεσης. Στο ψήφισμα του 2011 το Κοινοβούλιο ανέφερε τις ανησυχίες του για τα εργασιακά δικαιώματα στο Ουσμπεκιστάν αλλά και για τα πεπαλαιωμένα συστήματα αγροτικής συγκομιδής που χρειάζονται βελτίωση και αποτελούν ένα εμπόδιο για την κύρωση αυτού του πρωτοκόλλου. Όπως ακούσαμε και στην ακρόαση που έγινε μετά από το καλοκαίρι. Η Διεθνή Οργάνωση Εργασία εξέφρασε θετικά σχόλια για τι αλλαγέ στο Ουσβεκιστάν. Λέει ότι έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματα τη παιδική εργασία και μειώνεται συνέχεια η παιδική εργασία. Δυστυχώ εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο δρόμο να διατρέξουμε για να ξεπεραστεί το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας. Όπως μπορούμε να δούμε από την έκθεση του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας του 2015, το Ουσπεκιστάν έχει κάνει πολλές εκστασίες και έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να αυξήσει συνειδητοποίηση για τα θέματα εργασιακών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Το Ουσμπεκιστάν έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για τα θέματα αυτά. Το εμπόριο είναι σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη αυτών των σημαντικών εξελίξεων στο που έχει κάνει η χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια και έχει δείξει ότι έχει τη θέληση να αλλάξει τα πράγματα. Οι βελτιώσει ότι αφορά τη μεταρρύθμιση του αγροτικού συστήματο έχουν γίνει και σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα έχουν γίνει μείζονε βελτιώσει στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη σημασία της γεωστατικής ισορροπίας στην Κεντρική Ασία. Έχουμε χώρες οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν το κείμενο του ψηφίσματος φαίνεται ότι είναι καλό και εξισορροπημένο. Έχουμε κάποιες ανησυχίες για την παράγραφο 11 και την πρόταση για την ίχνη λασιμότητα, αλλά αυτά θα πρέπει να συζητηθούν τι επόμενες εβδομάδες και προσβλέπω στο να συνεργαστώ για την έκθεση αυτή. Αυτά είπε ο Χάνο. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος. Ο κ. Όμπερ Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και βλέπω ότι μετά από τις, ε, τις επιτροπές παρακολουθήσεως του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας φαίνεται να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό υποστήριζω αυτά που λέει η έκθεση. Τα είπε και ο Χάνου Τάκουλα στη δική του άποψη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα της ε, εργασίας, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της ε, μονοκαλλιέργειας στο Ουσπεκιστάν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντος με την κρίση παράστοκτων. Πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να βοηθήσει για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ώστε να οθήσει αυτή την περιοχή να προχωρήσει μια πιο αηφόρο μορφή ε, Η Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Κύριε Yes, uh, you, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Αρένα τις στις αρχές Σεπτεμβρίου συζητήσαμε το θέμα πιο εκτεταμένα και πάλι να πω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ουσπεκιστάν σε θέματα καταπολέμησης παιδικής εργασίας και ε, σε κάποιο βαθμό στο, σε ό,τι αφορά στην ε, καταναγκαστική εργασία Καλωσορίζουμε την συνεργασία ε, μεταξύ αρχών του Ουσβεκιστάν και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και πρέπει να βοηθήσουμε για να είναι εφικτή αυτή η συνεργασία. Χαιρόμαστε για την θετική έκβαση και ε, στην επιτόπου, στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη, είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα το κάνουμε σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και με την αντιπροσωπεία μας στο Ουσβεκιστάν και με χαρά θα ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όποτε κληθούμε ε, για τις εξελίξεις στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Η Μαρία, παρακαλώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι που πήραν το λόγο στηρίζουν τους προσανατολισμούς που προτείνω στην έκθεση και περιμένουν τις τροπολογίες σε σχέση και με το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε, γιατί το ψήφισμα θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες που οι Ουσβέκοι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν. Δηλαδή, ε, έχουμε τη συγκατάθεση, δίνουμε τη συγκατάθεση ε, για να με ότι αυτό που έχει γίνει είναι σημαντικό, αλλά τη δίνουμε επίσης ε, για να καλύψουν και το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής που τους μένει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. 16 Οκτωβρίου καταληκτική 17 Οκτωβρίου καταληκτική προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε το κείμενο στην Επιτροπή μας το Νοέμβριο και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια θα συζητηθεί το Δεκέμβριο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Με αυτά λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα για περίπου 7 λεπτά και μετά να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών.